benvenuti ai colleghi parlamentari e soprattutto. Λοιπόν, καλωσορίζω όλους τους συναδέλφους, καλωσορίζω κυρίω και τους ακροατές, τους φιλοξενούμενους που έχουν έρθει στην ακρόασή μα. Η ακρόαση αυτή διαιρείται σε δύο διαφορετικά πάνελ. Ε, εντάσσεται στα πλαίσια της έκθεσης Harbor για την ενιαία αγορά της τηλεπικοινωνίας. Γι' αυτό θα δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Χάρμπορ για να κάνει την παρουσίαση του θέματος και αμέσως μετά θα περάσουμε στις δύο διαφορετικές συζητήσεις, τα δύο διαφορετικά πάνελ θα προηγηθούν κάποιες σύντομες ανακοινώσεις από πλευράς ορισμένων προσκεκλημένων, θα ακολουθηθούν από ερωτήσεις και σχόλια από πλευράς των βουλευτών και στο τέλος θα δοθεί η τελική σύνθεση της συζήτησης, στο τέλος της δίωρης αυτής ακροάσεως από πλευράς του εισηγητή. Ξεκινάμε λοιπόν για να κερδίσουμε λίγο το χρόνο που χάσαμε μέχρι τώρα. Ο κ. Χάμπορ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητέ Αντιπρόεδρε, μιας και είμαι εισηγητής για το κομμάτι του θέματος που αφορά την ΙΝΚΟ, θα ήταν πιο ελεύθερο για μένα να πάρω μέρος στη συζήτηση αν εκχωρούσα την Προεδρία στον συνάδελφο. Δεν χρειάζεται μεγάλη εισαγωγή. Βλέπω εδώ τον κύριο Κρόιτσμαν, τον κύριο Έγκστρομ, και άλλους συναδέλφους και όδης εισηγητές. Ελπίζω ότι θα έρθει και η κυρία Μπαστός και άλλοι. Έχουμε ήδη συναντηθεί γύρω από αυτό το θέμα επανειλημμένα και είναι ασυνήθιστο να υπογραμμίζω ότι η έκθεσή μου έχει ήδη κυκλοφορήσει. Σε αυτήν την Επιτροπή συνήθως οργανώνουμε μία ακρόαση πριν ολοκληρωθεί η πρώτη έκθεση του εισηγητή αλλά λόγω της χρονικής πίεσης η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή που είναι η βιομηχανία ε, έχει ετοιμάσει το πακέτο που ονομάζεται Connecting Continents, δηλαδή συνδέοντας υπήρους και είναι διαθέσιμο και περιλαμβάνει και το δικό μου κομμάτι σε ένα πρώτο επίπεδο. Και αυτό είναι ασυνήθιστο. Θα οργανώσουμε μια συνάντηση με εμπειρογνώμονες και έχω προσκαλέσει και τους συναδέλφους να σχολιάσουν την έκθεσή μου. Πρώτα θα ακούσουμε όμως τις απόψεις των εμπειρογνωμόνων. Ελπίζω να σχολιάσουν τις προτάσεις μου και να ασκήσετε κριτική στις προτάσεις μου, γι' αυτό άλλωστε τις έχω κάνει. Πείτε μας αν είναι κάτι το θετικό Κάπου κάπου μπορεί κάποιες από τις προτάσεις μας να γίνονται δεκτές ευμενώς. Και μετά θα έχουμε ένα 20 λεπτό οι συνάδελφοι αν θέλουν να προσθέσουν και διαφορετικά σχόλια και σημεία ε, για να ορίσω κάπως τους όρους της συζήτησης. Η ευθύνη της Επιτροπής μας συνδέεται με τις προηγούμενες εργασίες μας. Ήμασταν υπεύθυνοι στο παρελθόν για, τις λεγόμενες, για την οδηγία για τις λεγόμενες ε, καθολικού τύπου υπηρεσίες. Αυτό είναι βασική μας ενασχόληση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ξεκίνησε την εποχή που η ενιαία αγορά ανήκε περισσότερο στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. και ενιαίας αγοράς. Εγώ τότε ήμουν εισηγητής για την βασική πρόταση σχετικά με το πακέτο Telecom, το οποίο είχε γίνει δεκτό το 2002 και μετά ήμουν εισηγητής πάλι όταν έγινε η αναθεώρηση του πακέτου αυτού το 2009. Είναι μια ιδιαίτερη, αν περίπτωση το να είναι βουλευτής εισηγητής κάποιος ο οποίος έχει εργαστεί με δύο διαδοχικούς επιτρόπους. Και θα ήθελα να πω ότι εξεπλάγει στα πλαίσια της δεύτερης διαδικασίας αναθεώρησης. Τώρα είμαι και για μια ακόμη φορά, για τρίτη φορά εισηγητής πάλι. Δεν ξέρω, ίσως λοιπόν να είμαι γνώστης ίσως και όχι τόσο, πάντως οι συνάδελφοι με, ε, μου ανέθεσαν τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα να εξετάσω δηλαδή τις προτινόμενες αλλαγές μεταρρυθμίσεις στα δικαιώματα των χρηστών. Η έκθεσή μου έχει εξετάσει αυτά τα οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την βελτίωση των δικαιωμάτων των χρηστών. Στα πιο πολλά συμφωνούμε, αλλά δεν συμφωνούμε με τον τρόπο που συνδέεται αυτό στα πλαίσια του νομοθετικού πακέτου. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο δημιουργεί μια κάποια σύγχυση βλέπουμε ότι 28 αρχές έχουν εφαρμόσει επιλεκτικά τέτοιου είδους τμήματα του πακέτου και βλέπουμε παράλληλα ότι οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί μέσω ακριβώς του κανονισμού μεγιστοποιούν την εναρμόνιση, αλλά ανερών από τις ρυθμιστικές αρχές την απαιτούμενη ευελιξία για τη διαχείριση μιας ευαίσθητης αγοράς. Αυτό το οποίο προσπαθήσαμε λοιπόν να κάνουμε είναι να επανεπαξεργαστούμε κάποιες από τις ιδέες που περιλαμβάνονται στην οδηγία για τα δικαιώματα των χρηστών και που καλούνται να εφαρμόσουν οι διαχειριστικές αρχές. Ένα άλλο θέμα στο οποίο μπορεί να διαφέρουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτεί να παρεμβαίνει σε επίπεδο ιδιαίτερος λεπτομεριακό σε σχέση με τα πράγματα. Εμείς διαφωνούμε με αυτό. Ήδη από το 2009 είχαμε πει ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Σώμα Εθνικών Δυθμιστικών Αρχών του τομέα των τηλεπικοινωνιών. Έχουμε αρχίσει να συνεργαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή έχουν αρχίσει οι πιέσεις μεταξύ των αρχών αυτών για να υπάρξουν αλλαγές και ναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συμβάλει προς την κατεύθυνση αυτή τη διακανονιστική λέγοντας ότι σε ορισμένες αγορές γύρω στις 10 δεν έχουν εφαρμοστεί οι προβλεπόμενες αλλαγές και στόχος μας είναι το υπάρχον ρυθμιστικό πλαίσιο να λειτουργήσει. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία όμως για να περιπλέξουμε το σύστημα, να συγκεντρώσουμε τις εξουσίες σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με επιλεκτικό τρόπο να ζητήσουμε την επιβολή των διακανονιστικών ρυθμίσεων. Συμφωνούν οι συνάδελφοι οι σκιώδεις με αυτό και γι' αυτό διαμορφώσαμε την πρότασή μας. Το θέμα αυτό που είναι πολιτικό θέμα δεν μειώνει την μεγάλη σημασία της εφαρμογής του πακέτου των δικαιωμάτων των Χριστών στις τηλεπικοινωνίες. Αυτό είναι το πρώτο τμήμα λοιπόν, το πρώτο κομμάτι της απογευματινής μας συνεδρίασης. Και θα θέλαμε να ακούσουμε σχόλια για τη βελτίωση των δικαιωμάτων των Χριστών, αν το πετύχαμε, αν κάναμε λιγότερα ή αν κάναμε περισσότερα από όσο έπρεπε. Το δεύτερο, και αφού συμφωνήσαμε ότι πρέπει να υπάρξει ένας κανονισμός, είναι να δούμε ποιες είναι, ποια είναι τα στοιχεία αυτής ε, της πρότασης σχετικά με την πρόσβαση των χρηστών, με θέματα ουδετερότητας του δικτύου, με τις ανησυχίες σχετικά με την net neutrality. Περνάμε σε ένα διαδίκτυο υψηλής χωρητικότητας, με πολλαπλές χρήσεις και εφαρμογές, με νέες υπηρεσίες μέσα από τα ίδια φάσματα. Και εδώ υπάρχουν περιθώρια για διακριτική μεταχείριση από πλευράς των εταιριών που ελέγχουν το δίκτυο και των παρόχων. Η ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό σε ό,τι κάνουν οι πολίτες και γνωρίζουμε ότι σε νομοθετικό επίπεδο όλο και περισσότερο ε, υπάρχει ενημέρωση των καταναλωτών με ετικέτες κτλ Τώρα πολλές φορές αντικαθίσταται αυτό από μια διεύθυνση στο διαδίκτυο στην ουσία και γι' αυτό θα πρέπει ακριβώς αυτή η ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο να γίνει αντικείμενο εγγύησης, επίσημης εγγύησης μέσα στην συγκεκριμένη αυτή πρόταση. Η συζήτηση είναι λοιπόν για τον τρόπο με τον οποίο θα το πετύχουμε αυτό, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος, χωρίς να μειώσουμε την καινοτομική διάθεση, ε, τη σύνδεση νέων μέσων και σε επίπεδο ασύρματης ε, και σε επίπεδο ενσύρματης επικοινωνίας. Όλο και περισσότεροι χρησιμοποιούν την ασύρματη επικοινωνία βέβαια, και το ευρύ φάσμα και αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αυτά. Και τώρα θα σταματήσω να ομιλώ και θα ακούσω τις απόψεις των εμπειρογνωμόνων και θα ζητήσω και από τους συναδέλφους να κάνουν σχόλια σε αυτά που θα ακούσουμε, γιατί όλα αυτά θα αντικατοπτριστούν στις επόμενες τροπολογίες που κατατεθούν στην πρότασή μου. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο πάνελ όπως ήδη ανέφερε ο Πρόεδρος, μετά κατά διάρκεια της συζητήσεως θα δώσω το λόγο και στους ε, συναδέλφους σκιώδης εισηγητές και μετά σε όλους τους συναδέλφους που θα ζητήσουν το λόγο, θέλουν να υποβάλουν ερωτήσεις ή θέλουν να τοποθετηθούν, να εκφράσουν απόψεις. Και ο Πρόεδρος θα τα λάβει όλα αυτά υπόψη του στη σύνταξη των ε, κειμένων του. Όπως γίνεται κανονικά σε τέτοιες ε, περιστάσεις. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ξεκινήσω δίνοντας το λόγο στον κύριο Πολ Ότον που είναι ο πρώτος εισηγητής που θα μιλήσει στο πρώτο τμήμα αυτής της ακρόασης. Λοιπόν, θα ζητούσα και από εκείνον και από τους άλλους αν έχουν την καλοσύνη την παρουσίασή τους να την περιορίσουν χρονικά σε ένα δεκάλεπτο που προβλέπετε ούτω ώστε να μπορούν να έχουν χρόνο να μιλήσουν και οι συνάδελφοι. Έχετε το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Πούλε Χάπτον είναι το όνομά μου. Και είμαι από το WITCH, από την Ένωση Καταναλωτών του Λονδίνου. Μιλώ βασικά εκφράζοντα άποψη του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά ο συνάδελφός μου θα μιλήσει αργότερα. Θα αναφερθεί σε διάφορε στοιχεία. Αυτά που θα πω ε, εκπροσωπούν ουσιαστικά την μεγαλύτερη, τα, μέλη της άλλης ε, ε, ένωσης καταναλωτών της Μπερ. Λοιπόν, βασικός στόχος της ψηφιακής ενίας αγοράς είναι αυτός που θέλω να αναφέρω και κυρίως τα δικαιώματα των καταναλωτών. Θεωρούμε ότι οι προσπάσεις που καταβάλλονται εκεί είναι ένα βήμα πρόοδου. Τα περισσότερα σχόλιά μου θα τα περιορίσω σε αυτό το κομμάτι της παρουσιάσεως. Για το γενικό πακέτο εμείς δεν θέλουμε να ξεχάσουμε την ανάγκη για ανταγωνισμό και για ενοποίηση. Τώρα τέθηκε κατά πόσο αυτό είναι το σωστό βήμα και όχημα για να πετύχουμε τους στόχους μας. Δεν ξέρουμε ποια είναι η απάντηση αυτό. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι στα πλαίσια του, της οδηγίας ή του σχετικού κανονισμού όπως αυτός υποστηρίζουμε την ελάχιστη εναρμόνιση. Και θέλουμε να βρούμε τρόπο να το πετύχουμε. Και αν μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος μέσω τροπολογιών που θα οδηγήσουν σε διαφορετικό νομοθέτημα είναι κάτι που το υποστηρίζουμε. Τώρα γι' αυτό θα συζητήσουμε τα διάφορα τμήματα. Υποστηρίζουμε το πνεύμα της πρότασης. Ταιριάζει με το περιβάλλον που τονώνει τον ανταγωνισμό. Δίνει δύναμη στον τομέα βοηθά τον κόσμο, βοηθά τους καταναλωτές, τους δίνει κάποια δύναμη, τους μαθαίνει πώς να έρχονται σε επαφή με τους παρόχους υπηρεσιών Άρα τους ενημερώνει τους ε, πολίτες πριν συνάψουν τη σύμβαση, όταν έχουν υπογράψει την ε, σύμβαση, πώς αλλάζουν πάροχο κλπ. Καλύπτονται όλες οι φάσεις. Υπάρχει μια ανησυχία ότι περιέχονται πολλά. Σαν αποτέλεσμα αυτού, ίσως θα υπάρξει κάποια μετακίνηση κόστους, σημαντική μάλλον. Πρέπει να δούμε κατά πόσο μετακυλίονται οι δαπάνες από ένα τομέα σε άλλον. Πρέπει να το εξετάσουμε αυτό. Ίσως γι' αυτό πρέπει να υπάρχει στο μέλλον δυνατότητα αναθεώρησης, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο των προτάσεων. Πριν αναφερθώ στις συγκεκριμένες προτάσεις του κανονισμού, να πω κάποια πράγματα όσον αφορά το πώς βλέπουμε εμείς τα ζητήματα αφορούς καταναλωτές στην αγορά. Θα τα ομαδοποιήσω σε τρεις, τα προβλήματα σε τρεις τομείς. Πρώτον, ενημέρωση και ο περίπλοκος χαρακτήρας του τομέα. Δεύτερον, ποιότητα υπηρεσιών. Τρίτον, η διαδικασία αλλαγής παρόχου. Πρώτος τομέας, πληροφορίες και περιπλοκότητα αυτών. στον τομέα των κινητών ο κόσμος ξέρει κάπως τις διάφορες έννοιες. Τα θέματα των λεπτών και τα διάφορα μηνυματάκια τα γνωρίζει ο κόσμος. Πιο δύσκολα τα πράγματα είναι όσον αφορά τα στοιχεία, τα δεδομένα. Έγινε έρευνα στον Ηνωμένο Βασίλειο, πολύ ενδιαφέρον. Από το Bill Monitor, μια οργάνωση. Και κατανοητές στον Ηνωμένο Βασίλειο πληρώνουν υπερ... παραπάνω περίπου κατά 6 δισεκατομμύρια το χρόνο στους λογαριασμούς τους. Είτε ε, μάλλον υποεκτιμώντας τον όγκο των δεδομένων που χρησιμοποιούν. Άρα ο περίπλοκος χαρακτήρα του τομέα δημιουργεί προβλήματα. Κυρίως όσον αφορά τη, μεταβίβαση, τη μετάδοση δεδομένων. Άλλαξαν και οι όροι. Όταν αλλάζουν οι όροι κατά τη διάρκεια της σύμβασης, εκεί επικεντρώσαμε τις προσπάθειες. Κάναμε μια εξετατή αρκετά επιτυχή στον Αμένο Θέλαμε ο κόσμο να απομακρυνθεί από συμβάσεις αν κατά τη διάρκεια της, του, σύμβασης ανεβούν οι τιμές. Μετά, δεύτερο τομέα, η ποιότητα των υπηρεσιών. Κάναμε έρευνα πέρσι τον Μάιο. Ρωτήσαμε τα μέλη μας. Θα κάνουν το ίδιο και φέτος. Ρωτήσαμε ποια είναι τα περισσότερα προβλήματα, τα μεγαλύτερα για την ευρυζωνική, 29% του κόσμου έλεγε ότι είναι αργές οι ευρυζωνικές περιπτήσεις. 18% πολύ συχνά ότι υπάρχουν διακοπές και 15% είπαν ότι δεν είχαν σύνδεση για ώρες ή για μέρες. Υπάρχουν κάποια προβλήματα λοιπόν. Στον, κινη... Στον τομέα των κινητών υπάρχουν κάποια προβλήματα, κυρίως αφορά την κάλυψη. Όλοι το καταλαβαίνουν ότι θα έχουν παντού κάλυψη δείχνουν κατανόηση. Αλλά στο σπίτι, άμα υπάρχει έλλειψη κάλυψη ή στον τόπο εργασία, εκεί υπάρχει πρόβλημα, ενοχλούνται. Και μετά το άλλο θέμα, το τρίτο, αλλαγή. Παρακολουθήσαμε τι έκαναν 5.000 μέλη μα. Του μιλήσαμε τον Μάρτιο και μετά τον Μάιο. Τον Μάρτιο έλεγαν ότι θα κάνουν αλλαγή παρόχου και τον Μάιο πήγαμε και του ρωτήσαμε να δούμε αν πράγματι άλλαξαν. Μόνο το 1 τρίτο εκείνων που είχε πρόθεση να αλλάξει το έκανε. Πολλοί λοιπόν παρετούνται από τη διαδικασία αλλαγή και θέλαμε να καταλάβουμε γιατί. Ο 34% του κόσμου είπε ότι παρετήθηκε διότι φοβόταν ότι κάτι θα πήγαινε στραβά με την αλλαγή. 32% είπαν ότι η διαδικασία ήταν δύσκολη. 12% είπαν ότι ο πάροχός τους τους έδωσε κίνητρα να μείνουν. Από πλευράς αντίληψης, πώς βλέπει ο κόσμος το το όλο θέμα υπάρχουν προβλήματα αλλαγή παρόχου. Και μετά άλλα θέματα που καλύπτει η οδηγία. Ε, το bundling, η ομαδοποίηση των υπηρεσιών, δημιουργία φρόχων και ή ε, πακέτων μάλλον υπηρεσιών. Είναι ένας λόγος που δεν θέλει να μετακινηθεί κάποιος. Και στον τομέα των κινητών το θέμα της ε, καρτούλας, της SIM και της αλλαγής αυτής που ίσως να πρέπει να πληρώσει για να αλλάξεις. Εκεί λοιπόν είδαμε ότι δημιουργούνται προβλήματα για του καταναλωτέ. Όσον αφορά τι προτάσει που έχουμε μπροστά μα, όπω είπα στην αρχή, είναι πρόσδεκτε. Ε, καλύπτουν ευρύ φάσμα. Όλη την πορεία που ακολουθεί ο καταναλωτή. Δεν έχω συγκεκριμένα σχόλια όσον αφορά τα σημεία που αναφέρονται στην ενημέρωση. Καλό το πακέτο των μέτρων που προτείνονται. Υποστηρίζουμε την πρώτα σύμφωνα με την οποία πρέπει να επιτρέπεται ο κόσμος να βάζει ανώτατο όριο εθελοντικά στη χρήση. Ερευνήσαμε και αυτό το θέμα τον περασμένο μήνα. Η έρευνα αυτή δείχνει περισσότερο τις προθέσεις των ανθρώπων παρά αυτό που έκαναν. 24% όμως είπαν ότι αυτό αν γινόταν θα το ενστερνιζόταν, αν είχαν τη δυνατότητα. Υποστηρίζουμε και το μέτρο για τη διάκριση των, των ε, των ε, περαστικών τηλεφωνημάτων για το Ηνωμένο Βασίλειο μάλλον, περαστικών, ε, μάλλον από το Ηνωμένο Βασίλειο σε άλλη χώρα. 9 πένες το λεπτό για ντόπιο τηλεφώνημα εσωτερικό και 23 για να τηλεφωνήσει κανείς, 23 πένες το λεπτό για να τηλεφωνήσει η Γαλλία και η Γερμανία. Η ποιότητα των υπηρεσιών. Κάναμε μια εκστρατεία αρχέ του έτου, για αυτό το θέμα και ο ρυθμιστικός μας φορέας επέτρεψε πρόωρο τερματισμό. Υποστηρίζουμε λοιπόν και αυτό και το εξάμεινο υποστηρίζουμε. Εξάμεινο μπορεί να θεωρηθεί από τη μια αυθαίρετο νούμερο. Έχει αυξηθεί η διάρκεια των συμβάσεων. Πολλοί έχουν τώρα 24 μήνη σύμβαση. Θέλουμε όμως θέλουν η σύμβαση να είναι αρκετά μεγάλη για να καλύπτει εκτόσεις ή το κόστος κινητών τηλεφώνων που δίνονται. Αλλά παρόλα αυτά θα ήταν λογικό να θέσουμε μικρότερο, μικρότερη χρονική κλίμακα όσον αφορά αυτό το θέμα και υποστηρίζουμε και τα μέτρα για το να ξεμπλοκάρουν οι μικρές καρτούλες οι SIM και να μεταφέρονται εύκολα και να γίνει εύκολη διαδικασία. Όσον αφορά την αλλαγή παρόχου, είπα ότι ο κόσμος παρετείται από αυτό από την πρόθεσή του παρετείται γιατί δυσκολεύεται με την όλη διαδικασία. Άρα πρέπει να γίνει πιο εύκολη διαδικασία. Υποστηρίζουμε το άρθρο 30 και το κινητό της μιας ημέρας Δεν ξέρουμε πριν να είναι βασική πρόταση, το υποστηρίζουμε όμως πρώτα απ' όλα. Πρέπει να υπάρχει συνέπεια στην προσέγγιση αν υπάρξει αλλαγή, όλοι πρέπει να την εφαρμόζουν παρομοίως. Αυτοί που έχουν τα σωστά κίνητρα θέλουμε να κάνουν την αλλαγή και να κερδίζουν. Και αυτοί που κερδίζουν περισσότερα, δηλαδή η εταιρεία προ οποία κινούνται οι περισσότεροι, να έχουν λόγους για να αποκτήσουν τα κέρδη από τη μετακίνηση αντίθετα με το να βασιστούμε στους χρήστες. Το πακέτο γενικά είναι καλό, καλύπτει τα περισσότερα ζητήματα που εντοπίσαμε, τα προβλήματα, μιλώντας στα μέλη μας και στο ευρύτερο κοινό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στον κύριο Κίπμεϊκ διευθυντής του Everything Everywhere. Τον παρακαλώ και αυτόν να τηρήσει το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Έχετε το λόγο. Um, <coughs> um, <coughs> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Απλά για να εξηγήσω κάπως uh, everything everywhere, τα πάντα παντού. Είμαστε ουσιαστικά για το EE, e, για το uh, την δυνατότητα συνεργασίας Orange και Deutsche Telekom ηλεκτρονικά. Δεν κάνω λόγο, δεν εκπροσωπώ οποιαδήποτε από τις δύο εταιρείες, ωστόσο λαμβάνω υπόψη τις απόψεις τους στα όσα θα εκθέσω αμέσως μετά. Έχω κάποιες διαφάνειες που θα τις ε, εξηγήσω και θα τις περάσουμε γοργά και θα δώσω κάποια στοιχεία αρχικά για το ΙΙ και την βιομηχανία της επιχειρήσης και θα κάνω κάποιες ουσιώδεις παρατηρήσεις επί της ουσίας ε, προτού πάμε στα περαιτέρω θέματα που πρέπει να συζητήσουμε σήμερα. Λοιπόν, στη συνέχεια δεν θα περάσω γραμμή με γραμμή όλα τα κείμενα των διαφανειών. Θα πω κάποια πράγματα για τις επιχειρήσεις οι επιχειρήσει κινητών, τηλεφωνία είναι πολύ ευκίνητε στην Ευρώπη. Υπάρχουν τέσσερι εταιρείε που δίνουν σκληρή μάχη για να έχουν συμβόλαια. Είναι ένταση κεφαλαίου επιχειρήσει με υψηλό βαθμό και υπάρχει και παγκόσμιο ανταγωνισμός όσον αφορά άλλες εταιρείε ανταγωνιστικές και φυσικά δεν έχουν όλες το ίδιο επίπεδο, δεν υπάρχουν για όλες το ίδιο επίπεδο το ρύθμισης ε, όπως για τις ε, ίδιες τις ε, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Και αυτό είναι στοιχείο σημαντικό και πρέπει να αποτελέσει μέρος που θα συνεξεταστεί τμήμα συνεξέτασης σε σχέση με τις επιχειρήσεις. Αν δει κανείς την επιστροφή κεφαλαίου τα κέρδη όσον αφορά τις ε, κινητές αυτές ε, επικοινωνίες ε, για τις επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν μεγάλα περιθώρια, δεν έχουν περιθώρια κέρδους. Είναι μια πολύ σκληρή μάχη που δίνουμε σε αυτά τα περιθώρια. Υπό αυτούς τους όρους να υπάρχει το σωστό ρυθμιστικό πλαίσιο είναι σαφές ότι έχει ζωτικότατη σημασία. Και έτσι όταν εξετάζουμε αυτό το κείμενο ως νομοθετικό κείμενο και πρέπει εδώ και να ξέρω ότι με υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχω καλούς φίλους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλω να τους προειδοποιήσω όμως ότι δεν είμαι μέγας οπαδός αυτού του νομοθετικού κειμένου το κλειδί είναι ότι οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση πρέπει να εξετάζεται με σαφή αυστηρά κριτήρια και να δούμε σε σχέση με αυτά τα κριτήρια και τις αρχές αυτής της διαφάνειας. Δεν θα επισέθω σε λεπτομέρειες, γιατί θέλω να επισέθω σε περαιτέρω λεπτομέρειες στη συνέχεια αυτή η διαφάνεια είναι κάπως δύσκολο ίσως να αναγνωστεί, αλλά ουσιαστικά τι κάνει κάπως μεροληπτικά εντός εισαγωγικών εξετάζει κάποια από τα κριτήρια και εξετάζει αν αυτό το κείμενο νομοθετικό ανταποκρίνεται σε αυτά τα κριτήρια. Θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ καλό νομοθετικό κείμενο, μια και στρέφεται και εντοπίζει σαφώς τα προβλήματα έλλειψης, για παράδειγμα, επενδύσεων σε αυτό το τομέα στην Ευρώπη και έχει και άλλα καλά στοιχεία. Παράδειγμα, θα μπορούσα να επιλέξω και άλλα προτερήματα, αλλά θα επιλέξω το συγκεκριμένο εξή <clears throat> για το πώς θα έπρεπε το spectrum φάσμα να εναρμονιστεί, να ρυθμιστεί. Και ο μεγαλύτερος βαθμός εναρμονισμού που θα έπρεπε σε αυτό το φάσμα, σε αυτό το εύρος σπέκτρουμ ε, να επιτευχθεί στην Ευρώπη. Εκείνο όμω που δεν μας αρέσει και είναι κλειδί ότι περικόπτονται, περιστέλλονται τα υφιστάμενα νομοθετικά μέσα. Και όχι επειδή πιστεύουμε ότι αυτό το πλαίσιο αυτών των νομοθετικών ρυθμίσεων που ο Μάκομ Χάρμπορ ω εισηγητής ε, είχε στενά συνδεθεί με αυτό, όχι επειδή αισθανόμαστε ότι είναι τέλειο δεν το θεωρούμε ως τέλειο. Είναι όμως αρκετά καλό και παρήχε ένα πολύ θα έλεγα ένα πλήρες ε, πλαίσιο στο οποίο θα μπορούσαν να λαμβάνονται οι αποφάσεις για τις επενδύσεις στην Ευρώπη. Ένα όμως από τα πράγματα που δεν μας αρέσουν σε σχέση με αυτές τις προτάσεις είναι ότι χρησιμοποιεί διαφορετικά νομοθετικά μέσα και εργαλεία για να αντιμετωπιστούν κάποια από τα ίδια όμως κοινά προβλήματα και έτσι υπονομεύονται κάποιοι από τους όρους που προηγούμενα υφίσταντο και μπορούσαμε μέσα αυτούς να λειτουργούμε ως πλαίσια. Λοιπόν, δεν θα επισέθω σε λεπτομέρειες και πάλι επ' αυτών, αλλά η παρατήρηση για τα στοιχεία που δίνουν αυτή την κατεύθυνση όπως τροποποιήθηκε από το Telecoms Framework, το πλαίσιο ε, για τις τηλεπικοινωνίες του 2002, όπως τροποποιήθηκε και μεταρρυθμίστηκε ε, το 2009, μεταξύ των κύρια εμπλεκόμενων όπως ε, ημών, υιοθετούμε και εγκρίνουμε σε μεγάλο βαθμό τις προτάσεις, πρέπει να πούμε, του εισηγητού, Malcolm Harbour να προσπαθήσουμε να επανεντάξουμε, να επανενσωματώσουμε αυτές τις ε, διαφορετικές νομοθετικές προτάσεις σε ένα ενιαίο πλαίσιο, ώστε να μην υπονομεύεται, α το πω έτσι, η γενική αρχή, να μην υπονομεύονται οι αρχές που ε, θα πρέπει να εμπνέουν αυτό το πλαίσιο. Θα πρέπει όμως να γίνει αυτό με ένα πιο προσεκτικό, πιο συνετό τρόπο από αυτόν που ε, είχε προαχθεί τους τελευταίους μήνες. Ω θέματα αρχή αυτά. Α υπησέλθω σε κάποια θέματα λεπτομεριακά. Πρώτα, όσον αφορά τον, την βάσεων μετά από εξάμηνη περίοδο, για παράδειγμα. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό θα αυξήσει τα κόστη και την περιπλοκότητα και θα καταστήσει ε, πιο περίπλοκα τα πράγματα. Θα απαιτεί μια αναδόμηση, αναδιάρθρωση συμβολέων ε, εγκάρσια όσον αφορά τις ε, υπηρεσίες, τα συμβόλαια και τις υπηρεσίες που παρέχονται. Καλοχαιρετίζουμε την, καλοδεχόμαστε την πρόταση του εισηγητή να αρθεί, να καταργηθεί αυτό. Όσον αφορά τους σωστούς όρους και όσον αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων μεταξύ των όσων παρέχονται και όσων έχουν υποσχεθεί και τελικά παρέχονται χαιρετίζουμε την τροπολογία του, Ευρω... του εισηγητού να ληφθεί υπόψη ο μέσος όρος, ένας μέσος όρος ε, ε, και καθώς θα γνωρίζετε για τις ταχύτητες, οι ταχύτητες κυμαίνονται και σε μεγάλο βαθμό και έτσι ένας μέσος όρος θα έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη, είναι πιο χρήσιμο. Η τροπολογία που προτείνει ο εισηγητής ε, όντας ε, ε, μία πρόοδος, ε, δεν είμαστε απόλυτα πεισμένοι για την αναγκαιότητα γιατί στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με τους κανόνες για την διαφήμιση και την παρουσίαση θεμάτων που θα έπρεπε να μπορούν να αντιμετωπίζονται μέσω μιας ρύθμισης και όχι μιας παρέμβασης. Για την αλλαγή συμβολέων, contract switching, όσον αφορά την ε, περίοδο για μία ημέρα για παρεοχή για παροχή υπηρεσιών πέρα από, πάνω από μία μέρα οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι σημαντικές ε, όχι τόσο μόνο η ταχύτητα δεν μας αρέσει η ιδέα ότι θα πρέπει κάποιοι να, λαμβάνουν μια, να μπορούν να λαμβάνουν μία απόφαση ε, αποχώρησης ή προσχώρησης μέσα σε μία ημέρα θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη την ρύθμιση αλλαγής που υφίσταται στην Ευρώπη και πολλές εταιρείες ε, στην Ευρώπη έχουν επενδύσει σε συστήματα τα οποία είναι λιγότερο ταχαία από αυτή τη ρύθμιση. Το κλειδί για τον καταναλωτή δεν είναι αν θα είναι μια μέρα, δύο μέρες, τρεις ή τέσσερις ημέρες αλλά θα είναι το αν αυτή η αλλαγή θα μπορεί να γίνει χωρίς να διακοπούν οι υπηρεσίες ε, που παρέχονται. Διότι το θέμα της διακοπής υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα δύσκολο, δημιουργεί ιδιαίτερες δυσχέρειες ε, για τους ε, χρήστες, για τους καταναλωτές και θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι πολλές εταιρείες έχουν επενδύσει μεγάλα κονδύλια στα υφιστάμενα συστήματα και το να μεταλλαχθούν αυτά τα συστήματα για να ανταποκριθούν στον όρο της μιας ημέρας δεν θα, είχε, δεν θα παγόταν ε, μεγάλο ε, κέρδος και ούτε θα έδινε τίποτα ως ε, κέρδος στους καταναλωτές. Τώρα, σε σχέση με τις διεθνείς κλήσεις και τα SMS, τα ηλεκτρονικά μηνύματα, δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο, εκτός από το να πω ότι θεωρούμε ότι είναι απόλυτα περιττή αυτή η παρέμβαση. Είναι μια πάρα πολύ ανταγωνιστική αγορά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην δική της προσέγγιση μια και απέρριψαν την ανάγκη στη, κατά το παρελθόν παρεμβάσεων ή επεμβάσεων στην αγορά, δεν υπάρχει κανένας λόγος που να δικαιολογεί μια τέτοιου είδους ε, ε, παρέμβαση. Αλλά από πλευράς της Κοινοβουλευτική Επιτροπής και τι προτάσει που έχουν κατατεθεί στη δική σας Κοινοβουλευτική Επιτροπή και την Επιτροπή Ήτρε, θα θέλαμε ε, να σα πούμε ότι θα το καλωσορίζαμε πάρα πολύ αν θα μπορούσε να καταργηθεί αυτό ε, έλεγχος όσον αφορά την ε, ε, κατανάλωση, έλεγχος της κατανάλωσης σε σχέση με τις ανάγκες που υφίστανται. Θα ήθελα να πω επ' αυτού τις δικτυωμένες υπηρεσίες ή τα πακέτα υπηρεσιών που δημιουργούνται από τις υπηρεσίες που παρέχονται από τις εταιρείε μας. Από κάποιες από αυτές παρέχονται ήδη αυτές οι υπηρεσίες η αναλογία όσον αφορά τα έσοδα εκτός αυτών των δικτύων που μειώθηκαν σημαντικά κατά τα τελευταία έτη υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα που συνδέονται με αυτό το θέμα. Αυτό που θα ήθελα να πεθάνω ως έκκληση είναι αν προχωρήσουμε προς αυτή την οδό ρυθμίζοντας τα πράγματα αντί να υπάρξει ε, ατομική δέσμευση α ατόμων, ε, ας το πω έτσι, και ε, σε σχέση με συγκεκριμένες υποχρεώσεις, θα έπρεπε να έχουμε δεσμοποίηση, δέσμες που θα μπορούσαν να, να ε, λειτουργήσουν. Ίσως αυτό θα ήταν το ευθετότερο. Απλά και μόνο θα ήθελα να, να, ολοκληρώσω, να ολοκληρώσω με κάποια άλλα θέματα. Πρώτον, πολλά από τα θέματα καταναλωτών που αναφέρθηκαν αναγνωρίζουμε ότι υφίστανται και δεν ε, ε, τα αμελούμε. Πρέπει να αντιμετωπιστούν και, αν πρέπει, και όταν πρέπει να αντιμετωπιστούν τότε υπό το πρίσμα του ανταγωνισμού και ο όρος ανταγωνισμός ίσως ε, μπορεί εδώ να μην δίνει την ε, απόλυτη λύση και θα πρέπει με σωστή στάθμιση, ορθή, σωστή συνετή στάθμιση να προχωρήσουμε. Και έτσι να δούμε ότι η ταχύτητα η οποία ε, ε, έχει υιοθετηθεί η επιτάχυνση δεν είναι ίσως η πιο ενδεδειγμένη σε σχέση με τη συνετότερη στάθμιση. Και ένα άλλο θέμα σε σχέση με αυτό το θέμα αρχής είναι να βελτιωθεί το πλαίσιο. Το πλαίσιο παρέχει, θα πρέπει να παρέχει την βεβαιότητα που έχουν ανάγκη μέσα σε αυτή να λειτουργούν οι χρήστες. Και αυτό είναι το κυριότερο θέμα. Έχουμε υποεπενδύσεις ε, σε σχέση με τον τομέα των τηλεπικοινωνιών, σε σχέση με την Άπο Ανατολή, τις χώρες της Άπο Ανατολής. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα θετικό, ασφαλές ε, επενδυτικό περιβάλλον και αυτό να μπορέσει να λειτουργήσει θετικά και ως κίνητρο. Και όλα αυτά, δεδομένων όλων αυτών, πρέπει έτσι να προχωρήσουμε, να αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα μεταξύ μεταξύ των κυριότερων εμπλεκόμενων για να μπορούν να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον ασφάλειας. Τελευταία μου παρατήρηση. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μια σωστή αξιολόγηση του τι θα σημαίνουν όλα αυτά και ως ε, πρώην πρόεδρος της ε, Ρυθμιστικής Επιτροπής πρέπει να αναγνωρίσουμε το ότι αυτό θα πρέπει να εμπλέκει τον νομοθέτη σε σχέση με το ρυθμιστικό έργο στην Ευρώπη με μια σε βάθος γνώση των πραγμάτων και σε λεπτομέρειες ρυθμίσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι συγκρατημένη θα έλεγα ε, ακολουθώντας αυτή την οδό. Και θα έπρεπε τα θέματα λεπτομέρειας ε, να αφήσει να οριμάσουν και να εξεταστούν ε, με τον πιο συνετό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικότερες αρχές. Και πάλι εδώ θα ήθελα να πω έναντι της Επιτροπής ότι αυτό το εγχείρημα, ας το πω έτσι, υπερβολικά πολύ εμπλέκεται στη ρύθμιση λεπτομεριών και υπερβολική ρύθμιση. Και αυτό δεν νομίζω ότι είναι θετικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Στην κυρία Μπράντελ ο λόγος από το Digital Europe. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας έτσι ώστε να κάνω την παρουσίαση της οργάνωσής μου. Η Ένωση Digital Europe τι είναι είναι η φωνή της ψηφιακής βιομηχανίας, όπως την ε, ονομάζουμε, 57 εταιρείες, 36 εμπορικοί εθνικοί σύλλογοι και 10.000 συνολικά επιχειρήσεις στον τομέα του IT στην Ευρώπη. Παροχής ε, ε, κατασκευαστές ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ελεγκτές και παροχή δικτύων κτλ. Όταν προσπαθούμε να αναλύσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις αρχές του 2013, εξεπλάγημεν γιατί μετά από πάρα πολλές συζητήσεις που είχαν οδηγήσει στο νομικό πλαίσιο του 2009, ε, είδαμε ότι άρχισαν να εφαρμόζονται στις περισσότερες χώρες οι προτάσεις αυτές και ξαφνικά βλέπουμε μια νέα πρόταση για ένα νέο κανονισμό ε, και αυτό είναι κάτι το οποίο μας προκάλεσε μια κάποια έκπληξη. Βλέποντας τις λεπτομέρειες της συγκεκριμένης πρότασης είδαμε ότι ο στόχος είναι κάτι με το οποίο προφανώς συμφωνούμε, να δημιουργηθεί δηλαδή μια ουσιαστική ψηφική αγορά για τις τηλεπικοινωνίες είναι κάτι το καλοδεχόμενο. Ταυτόχρονα είδαμε ότι υπάρχει λόγος για τροπολόγηση των κανόνων οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ισχύ, αλλά πιστέψαμε ότι υπήρχε, ε, θα έλεγα, πιστεύαμε τουλάχιστον ότι υπήρχε ένα σύστημα απελευθέρωσης της αγοράς και με τους νέους κανόνες είδαμε ότι δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε τους στόχους αυτής της φιλελευθεροποίησης. Εμείς σαν ένωση που εκπροσωπούμε τη συγκεκριμένη βιομηχανική δραστηριότητα από πλευράς κατασκευαστών και παρόχων ε, υπηρεσιών, Θέλουμε να κάνουμε ό,τι γίνεται για να βελτιώσουμε τις επενδύσεις στον τομέα της δραστηριότητάς μας ε, και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ. και θα πρέπει να μην πάρουμε καμία απόφαση η οποία μπορεί να δημιουργήσει θέμα ή πρόβλημα στον επενδυτικό τομέα. Και αυτό παρακαλώ να το λάβετε υπόψη σας. Ταυτόχρονα θα έλεγα ότι οι βασικές μας ανησυχίες και τα βασικά θέματα είναι θέματα στα οποία δεν εμπλέκεστε άμεσα η εναρμόνιση της χρήσεως του εύρους που χρησιμοποιείται η κατανομή και κάποιοι άλλοι τεχνικοί κανόνες σχετικά με την δημιουργία αυτόνομων τοπικών δικτύων. Αυτά είναι θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν. Βλέπουμε ότι τέτοιου είδους προτάσεις θα μπορούσαν να είναι γενικότερα χρήσιμες. Ταυτόχρονα εμείς οι ίδιοι στη δική μας ανάλυση ασχοληθήκαμε με τις προβλέψεις με το θέμα της ποιοτικής παροχής προϊόντων, προϊόντων ποιότητας δηλαδή, και αυτό είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει άμεσα. Τέθηκαν και τα θέματα γύρω από τη λεγόμενη ουδετερότητα του διαδικτύου και το λεγόμενο ανοιχτό διαθέσιμο διαδίκτυο. Και εδώ πιστεύουμε ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε οτιδήποτε θα βελτιώσει την πρόσβαση στο διαδίκτυο και θα μας δώσει τη δυνατότητα για μεγαλύτερη νομική ευκρίνεια σχετικά με την διαχείριση, αν θέλετε, της κυκλοφορίας στο διαδίκτυο. Εδώ κάποιες ρυθμίσεις μπορεί να είναι λογικές και τεκμηριωμένες. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να οδηγήσουν σε αυτό το οποίο είπα στην αρχή, δηλαδή την ροή επενδύσεων στον τομέα, και αυτός είναι ο βασικός μας στόχος. Συνεπώς από πλευράς των, βιομηχανών, των βιομηχανικών εταιριών και των εταιριών παρόχων μπορούμε να υποστηρίξουμε αρκετά θέματα. Κάποια άλλα θέματα πρέπει να συζητήσουμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια Βασικός στόχο όμως είναι να καταστήσουμε τις προτάσεις αυτές συμβατές με την υπάρχουσα ήδη και λειτουργούσα νομοθεσία. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στη συζήτηση του ζητήματος. Στην πρώτη ακρόαση θα δώσω το λόγο αρχικά στους σκιώδεις εισηγητές και μετά προφανώς σε όλους τους συναδέλφους που θα το ζητήσουν. Δεν βλέπω τη συνάδελφο Μπάστος. Πάμε στους σοσιαλιστές. Η συνάδελφος Βεγνιού έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μιλάει εκτός μικροφώνου, δεν την ακούμε καλά δυστυχώς. Euh, Ευχαριστώ αυτούς που πήραν το λόγο. Για αυτό το θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε από σωστή διαπίστωση. Δεν είμαι καθόλου πεπισμένη όμως ότι βρίσκει τις σωστές απαντήσεις. Κυρίως όσον αφορά ε, το τέλος περιαγωγής. Κάποιος αναφέρθηκε στις συμβάσεις, εξάμηνες. Πρέπει να εξετάσουμε αυτή τη δήλωση, αντίθετα από το Μάλκομ θα πρέπει να υπάρχει επιλογή μεταξύ εξάμεινου και ενός έτους δύο ετών. Διότι διαφέρει από χώρα σε χώρα η κατάσταση. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για εναρμόνιση μέγιστη. Αναφέρθηκε μέγιστη εναρμόνιση. Δεν είμαι σίγουρη ότι προς αυτή θα πρέπει να κινηθούμε. Χρειάζεται ευελιξία σε επίπεδο κρατών. Στο Βέλγιο ένα συμβόλο εξάμεινο μπορεί να είναι ικανοποιητικό για το βέρο καταναλωτή. Στη Γαλλία βλέποντας τα στατιστικά στοιχεία πολλοί προτιμούν να μείνουν ένα ή δύο χρόνια με τον ίδιο πάροχο διότι τους δίνουν ε, κάποιες τιμές ειδικέ για κάποια συσκευή ε, ή τους προσφέρουν πολύ ενδιαφέρουσες ε, τιμές για συμβάσεις. Έχουν προσφορές. Νομίζω ότι το βασικό οικονομικό και μηχανικό διακύβευμα είναι οι επενδύσεις. Εκεί οι δημόσιοι φορείς ε, έχουν μειώσει σημαντικά τις πιστώσεις και αυτό το καταγγέλλω. Πρέπει να δούμε και ίσως μετά το συζητούμε αυτό, στο δεύτερο μέρος, να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε ισορροπία. Στο πακέτο αυτό βλέπετε υπάρχει το πακέτο των καταναλωτών και πρέπει να υπερασπιστούμε ε, όσο το δυνατόν ε, τους καταναλωτές και να προχωρήσουμε στη μεγαλύτερη δυνατή ευρωπαϊκή εναρμόνιση, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε τι γίνεται όσον αφορά τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Πώς μπορούμε να πετύχουμε την ισορροπία. Δεν θα πρέπει εκ νέου μέσω επενδύσεων μειωμένων ή κακού μερισμού των επενδύσεων να καταλήξουμε σε κατακαιρματισμό εδαφικό και κοινωνικό. Και όσον αφορά την ουδετερότητα του δικτύου θα το κουβεντιάσουμε, έχουμε πολλά να πούμε, κυρίως όσον αφορά την υποχρέωση διαφάνειας θα το αναφέρουμε μετά αυτό. Γι' αυτό είχα προβλέψει να πάρω το λόγο μετά για αυτά τα ζητήματα. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ Μπερναντέτ, συνάδελφε Κρόιτσμαν. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να σκεφτούμε πώς αυτή, τη σχηνοβασία, την ακροβασία θα την πετύχουμε μεταξύ ενός πολύ φιλοκαταναλωτικού καθεστώτος παράδειγμα δυνατότητα καταγγελίας μιας, ενός συμβολέου ε, σε ένα εξάμεινο και από την άλλη πλευρά να διασφαλίσουμε τις επενδύσεις από τις επιχειρήσεις όπως απαιτείται. Και ξεκινάμε τώρα με ένα νέο καθεστώς ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση απαιτούμε από τους παρόχους υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών πάντα να μας, να ε, θέτουν στη διάθεσή μας ένα ταχύτερο διαδίκτυο και έχουμε ήδη ταχύτατο ε, ε, διαδίκτυο, αλλά πόρο απέχουμε από την ε, παντελώς επιβολή του παντού. Απ' την άλλη πλευρά πρέπει να υπάρξουν επενδύσεις και χρόνος για αυτές τις επενδύσεις. Δεν είναι δυνατόν με μικρές, μικρής διάρκειας συμβόλαια να υπάρξει η ασφάλεια επενδύσεων, ώστε να μπορούν να αντληθούν εκείνα τα κεφάλαια και να επενδυθούν όπως απαιτείται. Γι' αυτό πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά τα πράγματα και να μεριμνήσουμε σε βάθος και συνετά να ρυθμίσουμε και όχι βιαστικά ελαφρά την καρδία. Να δούμε τι είναι εφικτό σε αυτή την νομοθετική περίοδο. Και όλα όσα είπα, είπε ο Μάκομ Χάρμπορ στην έναρξη αυτής της συνεδρίασης θα υποστηρίζουμε. Να προσπαθήσουμε να βρούμε μία πορεία όχι με βιαστικό τρόπο, όχι βιαστικά και ή μετά να υπάρξουν δισταγμοί από τα κράτη-μέλη ή να τα απορρίψουν τα κράτη-μέλη, να δούμε τι είναι εφικτό και μπορεί να γίνει σε αυτή την περίοδο. Και φυσικά για τα συμβόλαια αν ένα συμβόλαιο για 12 ας το πούμε έτσι περίοδο συνάπτεται και μετά υπάρχει ένας μήνας ε, περίοδος για να καταγγελθεί δεν θα είχαμε πρόβλημα να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή ενιαία εσωτερική αγορά αλλά ας μην έχουμε αυταπάτες. Θα πληρώσει ο καταναλωτής στο τέλος. Οι καταναλωτές θα πληρώνουν. Αν δεν υπάρχουν τέλη περιαγωγής πια, τότε οι επιχειρήσεις ε, ε, τηλεπικοινωνιών θα πρέπει να, όταν χρησιμοποιούνται υπηρεσίες ε, σε άλλη χώρα να πληρώνουν τα κόστη. και ποιος θα τα πληρώνει στο τέλος για να υποφελείται ο καταναλωτής. Να τα σκεφτούμε σε βάθος λοιπόν όλα τι μπορεί να γίνουν και τι είναι εφικτά και να μην πάμε βιαστικά, να αφήσουμε αυτά τα οποία είναι ανέφικτα για άλλη χρονική στιγμή και να θέσουμε ένα πλαίσιο με τέτοιο τρόπο ώστε όλα αυτά τα οποία εμείς επιθυμούμε να έχουμε δηλαδή να διασφαλίσουμε επενδύσεις στις υποδομές να τα πετύχουμε ώστε να υπάρχει δυνατότητα να έχουμε ταχύ διαδίκτυο στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Συνάδελφε Έκστρομ, έχετε το λόγο κύριε Έκστρομ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το θέμα της ουδετερότητας του δικτύου είναι ίσως το πιο σημαντικό για μένα θέμα του κανονισμού. Ο, ο λόγος για το, γιατί το λέω αυτό είναι ότι είναι ο μοναδικός τρόπος που μακροπρόθεσμα οι καταναλωτές θα έχουν καινοτομία και καλές συνθήκες είναι ο ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός είναι απαραίτητος και σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών από τους παρόχους και σε αυτό το πλαίσιο δυστυχώς ε, τα βραχυπρόθεσμα συμφέροντα της βιομηχανίας των τηλεπικοινωνιών αντίκυνται ε, στα συμφέροντα των καταναλωτών. Τις τελευταίες εβδομάδες συναντήθηκα με λόμπις από διάφορες επιχειρήσεις του διαδικτύου. Βασικά όλες λένε περίπου το ίδιο πράγμα, ότι θέλουν να εξειδικεύσουν τις υπηρεσίες τους και να καινοτομήσουν. Και όλες αυτές προσπάθησαν να με πείσουν ότι το διαδίκτυο δεν είναι αυτή τη στιγμή αρκετά ικανό για βίντεο, για παροχή βίντεο και γι' αυτό η τηλεόραση και το βίντεο πρέπει να παρέχεται μέσα από εξειδικευμένες υπηρεσίες. Ένας από αυτούς, μία από αυτές τις εταιρείες προσπάθησε να με πείσει για το αντίθετο αυτού που συμβαίνει εκεί που είμαι, ότι στο διαδίκτυο μπορεί κανείς να δει εύκολα βίντεο. Και νομίζω ότι το 90% του όγκου ε, που κινείται στο διαδίκτυο είναι τα βίντεο. Παρ' όλα αυτά η εταιρεία προσπάθησε να με πείσει ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο βίντεο από τη μία και την διαδικτυακή τηλεόραση από την άλλη και απέτυχε στην προσπάθειά του αυτή. Αυτό το οποίο επιθυμούν είναι οι εξειδικευμένες υπηρεσίες μέσα από τις οποίες θα, θα ορίσουν αυτές το παιχνίδι και αυτές θα αποφασίσουν αν κάποιος άλλος παροχέας θα έχει την δυνατότητα, θα έχει την άδεια να παρέχει υπηρεσίες στην ευρωπαϊκή αγορά και το τι θα πρέπει να πληρώσει στη συγκεκριμένη περίπτωση προς τον κύριο παροχέα. Ανησύχησα λοιπόν, αλλά δεν εξεπλάγει καθόλου από αυτού του είδους τα επιχειρήματα και από τους ε, εκπροσώπους της συνεργασίας Deutsche Telekom και Orange, που είναι δύο κυρίαρχα ολιγοπόλια τα οποία ελέγχουν την κυκλοφορία στο διαδίκτυο. Όταν αναφέρεται κανείς στο πώς η βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών θέλει στο μέλλον να αναπτυχθεί και θέλει να περάσει σε καινοτομικές προσφορές, λένε αυτά τα οποία θέλω εγώ να αποφύγουμε. Όλες οι επιχειρήσεις μέχρι τώρα στην Ευρώπη, όπως έχει συμβεί περίπου μέχρι τώρα, πρέπει να έχουν πρόσβαση στο, στο διαδίκτυο με προβλέψιμους όρους. Όμως η Orange και η Deutsche Telekom ε, θα θέλουν να είναι αυτοί που θα επιλέγουν το ποιος θα χρησιμοποιεί, το ποιος θα κερδίζει τη δυνατότητα χρήσης του διαδικτυακού φάσματος και ποιος όχι. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τα συμφέροντα, τα βραχυπρόθεσμα της βιομηχανίας των τηλεπικοινωνιών σε απόλυτη αντίθεση με τα συμφέροντα των αναγκών της εσωτερικής αγοράς και ε, των καταναλωτών. Ταυτόχρονα, όταν αναφέρεται κανείς στο ότι οι τηλεπικοινωνίες ελέγχονται στο κομμάτι το οποίο κανονικά θα έπρεπε να ελέγχονται στο κομμάτι το οποίο αφορά τις βασικές επικοινωνίες καθολικού χαρακτήρα. Εδώ πράγματι υπάρχουν κάποιες καταστάσεις οι οποίες αποτελούν απόκληση από τον κανόνα. Αν στην Deutsche Telekom της επιτρέψουμε σαν παράδειγμα να δημιουργήσει τις δικές της προσβάσεις σε κάποια δίκτυα και ταυτόχρονα να ε, ρίξει και να οδηγήσει όλους τους άλλους ε, παρόχους σε αργά συστήματα, τότε προφανές είναι ότι θα αποκτήσει μια ανταγωνιστική θέση υπέροχη εις βάρος των καταναλωτών. Συμφωνώ λοιπόν με κάποιες από τις γενικές παρατηρήσεις έκανε ο κύριος Χάρμπορ προηγουμένως Υπάρχει ένα πακέτο της Επιτροπής το οποίο συνολικά ε, έρχεται στο τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου αλλά και νωρίς σε επίπεδο επεξεργασίας. Αυτά που λέει η Επιτροπή τώρα για την ουδετερότητα του δικτύου δεν είναι λάθος αλλά δυστυχώς δημιουργείται μια τεράστια τρύπα στην αγορά, οι εξειδικευμένες υπηρεσίες, κάτι το οποίο θα επιτρέψει στους παρόχους να ευνοήσουν τις δικές τους υπηρεσίες ή τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι διατεθειμένες να πληρώσουν επιπλέον, κάτι το οποίο θα δημιουργήσει μια αβεβαιότητα και για τους μικρότερους επιχειρηματίες και κυρίως για τους χρήστες και καταναλωτές και όχι βέβαια για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Πρέπει λοιπόν πάρα πολύ σοβαρά να εξετάσουμε το θέμα των εξειδικευμένων υπηρεσιών. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να μετατρέψουμε τη συγκεκριμένη περίπτωση σε κάτι το οποίο θα βλάψει την εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Στίβαν ζήτησε το λόγο. Ή συνάδελφος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους ομιλητές μας και τους κοιόδης. Γιατί βρισκόμαστε εδώ, δεν έχουμε ενιαία αγορά. Διερωτώ με τι συζητάμε στις τηλεπικοινωνίες. Και γι' αυτό έχουμε την πρόταση. Εγώ θεωρούσα ότι η ιδέα της ενίας αγοράς ήταν αντί να έχεις 28 ομάδες ε, κανόνων, να έχεις έναν, ε, μία ομάδα κανόνων. Δεν ακούω τίποτα για το φέτσκιν τη αγορά. Ακούω πολύ αρνητική προσέγγιση, πολύ αρνητικά σχόλια, αρνητική διάθεση και αυτό με προβληματίζει. Για την περιαγωγή ε, πιστεύω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν αποκλίνουσε απόψει. Δεν πρέπει να το δυναμώσουμε. Αυτό που είπατε για τα δεδομένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και σαν κάποιο που προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το κινητό του τηλέφωνο και να δει ότι το έχουν, έχει τελειώσει το ότι δεν δουλεύουν τα δεδομένα και το Wi-Fi δεν δουλεύει στο κοινοβούλιο, δημιουργήθηκε κρίση. Ε, βλέπετε πόσο σημαντικές είναι οι υπηρεσίες αυτές στην καθημερινή μας ζωή και εδώ στο κοινοβούλιο. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω και για τον κύριο που αναφέθηκε στα δεδομένα και, και τον άλλο κύριο που μίλησε. Οι πελάτες, οι πελάτες σας τι σκέφτονται για τις ανάγκες τους σε δεδομένα διότι θα αυξηθούν οι ανάγκες. Είναι σημαντικό λοιπόν να πετύχουμε σωστή λύση. Το ότι δεν θέλετε ρύθμιση. Για να είμαστε ρεαλιστές, χρειαζόμαστε πλαίσια, τρόπους για τη δημιουργία βεβαιότητας και έτσι επενδύσεις. Με ενδιαφέρει πολύ η πλευρά του ανταγωνισμού, γιατί θεωρούσα ότι ο τομέας των τηλεπικοινωνιών σημαίνει ότι χρειάζονται επενδύσεις Πρέπει να επενδύουν εταιρείε για να είναι ανταγωνιστικέ και αυτέ οι επενδύσει πρέπει να απευθύνονται προς τους καλύτερους δυνατούς στόχους, προς όφελος των αναγκών των ε, καταναλωτών και για κάλυψη έναντι εξελίξεων μελλοντικών στην τεχνολογία. Για τα δεδομένα θέλω να ακούσω περισσότερα. Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που δεν υπάρχουν επενδύσεις. Προσπαθώ να το συμπεράνω και όσον αφορά το θέμα της ιδιωτερότητας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό Πολύ λίγοι γνωρίζουν πως σημαντική είναι αυτή η ιδιωτερότητα Είναι σημαντικό εμείς εδώ να πετύχουμε σωστή λύση. τέλος για, για τα συμβόλαια, σημαντικό ζήτημα για τους πελάτες Όλοι οι καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ε, πλαισιώνονται από δίκαιους κανόνε και όρους Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για να το πετύχουμε αυτό οι πελάτες και οι καταναλωτές να μπουν στο σωστό πλαίσιο, να μπορούν να απολαύσουν τα προσφερόμενα. Αυτοί οι όρη και που δεν ξέρει ο κόσμος ότι ανεβαίνουν τιμές και όταν θέλουν να αλλάξουν ε, υπάρχει κρυμμένο κόστος που δεν το ξέρουν. Αυτό είναι άδικο. Πρέπει να είναι δίκαιο το σύστημα. Αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε και θέλουμε να το υπογραμμίσουμε αυτό και να το τονίσουμε περισσότερο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλή τύχη. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος ο κ. Χάρμπορ ζήτησε το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον αυτά τα οποία ανέφεραν οι συνάδελφοι. Και κάποια σημεία θα ήθελα να αναφέρω και εγώ. Ιδιαίτερα για ένα ή δύο από τα θέματα λεπτομέρειας. Θα πρέπει να αναφέρουμε και ούτως ή άλλως υστερότερα κάποια άλλα. Θα περιοριστώ στα σχόλια που θα κάνω τώρα και μετά θα κάνω τα υπόλοιπα να πω σε σχέση με τα ωφέλη για τους καταναλωτές. Θα έλεγα και θα το ισχυριζόμουν αυτό, αλλά θέλω να ενισχύσω την παρέμβαση του προλαλήσαντος. Πιστεύω ότι το εφιστάμενο πλαίσιο εξυπηρέτησε πολύ θετικά τους καταναλωτές από το 2002. Εξελίχθηκε σταδιακά σταδιακά και έγιναν πολύ πιο ανταγωνιστικές οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών και οι τιμές μειώθηκαν. Ας μην το επανεκτιμούμε μη το υποεκτιμούμε, θα πρέπει πραγματικά να γίνουν και περισσότερα. Η δική μας κοινοβουλευτική ομάδα, η δική μας ε, κοινοβουλευτική επιτροπή ήταν εκείνη που έκανε την προσπάθεια να υπάρξουν όρια και να ε, προχωρήσουμε μέσα από τις σωστές διαδικασίες. Να τονίσω το εξής, τα όσα εγώ έχω αναφέρει δεν αλλάζουν τόσο σε σχέση με τη σημερινή πρόταση. Τι λέει η πρόταση, ότι μια συμφωνία που θα πρέπει να αναφέρει έναν αριθμό, έναν αριθμό για, που θα μπορεί να, ε, να καταλήξει σε, μέχρι σε μια συγκεκριμένη μέρα σε σχέση με το συμβόλαιο. Θα μας ενδιαφέρει να γνωρίζουμε αν ε, θα μπορούν οι, επιχει, οι επιχειρήσεις πάροχοι υπηρεσιών να έχουν δυσκολίες να προσαρμοστούν στους σημερινούς κανονισμούς ή όχι. Αλλά ανταποκρινόμενος στα σημεία τα οποία αναφέρθηκαν προηγούμενα, αν είναι ενδεδειγμένο να επιβάλλουμε κάποιους όρους ε, ή να επιβάλλουμε ρυθμίσεις ε, θα έπρεπε να πούμε ότι οι εμπλεκόμενοι που είναι υπεύθυνοι να ε, παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες θα πρέπει να είναι εκείνοι που θα είναι αρμόδιοι και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε σχέση με τις ρυθμίσεις ή απόψεις αυτές. Εγώ σε σχέση με την μικροδιαχείριση και μικρολεπτομέρειες στις οποίες εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπα ότι δεν πρέπει να επιβάλλονται ρυθμίσεις Ακόμα και όταν έχουμε λεπτομέρειες όσον αφορά τη μεταφορά μιας διεύθυνσης για παράδειγμα. Ε, αυτά είναι θέματα τα οποία δεν πρέπει να επιβάλλουμε σε σχέση με τις ε, ρυθμίσεις ε, και λεπτομέρειες. Γι' αυτό έχουμε ένα αποκεντρωμένο πρότυπο και όχι ένα κεντρικά σχεδιαζόμενο πρότυπο. Τώρα, σε σχέση με τις εξαμηνιές συμβάσεις ή συμβόλαια, εργαστήκαμε σκληρά να διασφαλίσουμε ότι θα έχουν πρόσβαση, θα έχουν δυνατότητες να αποχωρήσουν από ένα συμβόλαιο οι καταναλωτές αν αλλάζουν κάποιοι όροι. Αυτό θα έπρεπε να υλοποιείται με επιτυχία. Να μπορούν να επιβάλλονται οι όροι αυτοί σε σχέση με τα όσα προβλέπονται. Επίσης υπάρχουν διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες καταναλωτές έχουν υπόψη τους όρους και τις, πρέπει να έχουν υπόψη τους όρους και τις διατάξεις υπό τις, τους οποίους θα λειτουργεί το συμβόλαιό τους. Δεν πρέπει να υπάρχει αβεβαιότητα. Αν μετά από έξι μήνες για παράδειγμα ούτως ή άλλως λύγει ένα συμβόλαιο νομίζω ότι ούτως ή άλλως ε, παρέχουμε πάρα πολύ περίπλοκους όρους και διατάξεις για τους καταναλωτές. Οι βασικές διασφαλίσεις πρέπει να δίδονται ούτως ή άλλως. Η κύρια ανησυχία όμως που έχω είναι ότι θα υπάρχουν κάποιοι πάροχοι υπηρεσιών που θα επιβάλλουν και πριν για να τερματίζεται ε, ένα επρόσθετο ποσό το οποίο θα καταβάλλεται για να τερματίζεται ένα συμβόλαιο. Και αυτό θα είναι ένα αντικίνητρο στο να αλλάζει κανείς σύμβαση αν το επιθυμεί. Και πρέπει να το εξετάσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η συνάδελφος Τούν. Τελευταία παρέμβαση. Sorry, I was a little... Συγγνώμη, κάπως καθυστέρησα να προσέρθω. Ε, για την πρόταση της κυρίας Πιλάρ de και που θα έπρεπε να τα δούμε τα πράγματα. Κατάργηση δηλαδή των ε, επιπρόσθετων τελών που θα επιβάλλονται. Και ένα επιπρόσθετο θέμα, πρόσθετα σε αυτό, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ισοδίκαιο πλαίσιο για τη λειτουργία των εταιριών τηλεπικοινωνιών, δίκαιο για τους καταναλωτές, ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, πάυση της ε, ίσπραξης τελών για την ε, εκπνοή, για την λήξη ενός συμβολέου ή την καταγγελία μιας σύμβασης από πλευράς των καταναλωτών. Αυτό είναι κάτι το οποίο επανειλημμένα έχει προταθεί και την υποστηρίζουμε την κυρία Πιλάντε Καστίγιο σε αυτό το αίτημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πάμε στο δεύτερο μέρος της ακρόασής μας τώρα. Όμως οι ομιλητές ήθελα να ρωτήσω μήπως έχουν πρόθεση να απαντήσουν στις ερωτήσεις που τους ε, ετέθησαν. Το πολύ δύο λεπτά. Ο καθένας. Θα σας δώσω το λόγο με τη σειρά που πήρατε το λόγο πριν. Πρώτα ο κ. Χάουτον και μετά ακολουθούν οι υπόλοιποι. Προφανώς αν δεν έχετε τίποτα να δώσετε σαν απάντηση δεν θα, θυμώ, δεν θα θυμώσουμε μαζί σας ο κ. Χάουτον. Ευχαριστώ. Θα ήθελα σε κάποια από τα σημεία που ακούστηκα να σταθώ για τα δεδομένα. Νομίζω ότι το θέμα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το πιο καινούριο και το πιο περίπλοκο στις αγορές που μπορεί να κάνει ο καταναλωτής. Έχει μάθει ο καταναλωτής να πληρώνει, να χρεώνεται με λεπτά, ε, με, τα SMS φυσικά και το μέγεθός τους. Τώρα με τα δεδομένα είναι κάτι το σχετικά καινούριο, ο κόσμος τα χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο και για να κατεβάζει βίντεο κτλ. Και δεν είμαι βέβαιος ότι οι γνώσεις και οι προσδοκίες που υπάρχουν ε, αν είναι αντίστοιχες με την πραγματικότητα. Πολλοί κόσμος ίσως ε, να πέφτει σε λάθη, να κάνει λάθη. Και να υπάρχει πρόβλημα σχετικά με το κόστος το οποίο μπορεί να είναι πάρα πολύ υψηλό για την απαιτούμενη ισορροπία, για το τι πρέπει να περιλαμβάνει ο κανονισμός αυτός και τι δεν πρέπει να περιλαμβάνει. Ακούσαμε αυτά τα οποία είπατε σε σχέση με τις ανάγκες που υπάρχουν. Υπάρχουν πάρα πολλά τεχνικά θέματα βέβαια, η ε, περίπλοκα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν σε σχέση με την ταχύτητα μεταφοράς κτλ. Υπάρχουν επίσης κάποια άλλα θέματα τα οποία άπτονται του λογαριασμού των καταναλωτών όπως το τρόπος με τον οποίο θα ξεκινά η κατανάλωση ή όχι. Και θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα στο σωστό επίπεδο έτσι ώστε ό,τι χρειάζεται να γίνει να γίνεται στην κατάλληλη φάση. Ευχαριστώ λέει ο κ. Χιούτον. Ευχαριστώ. Κύριος Κίπε Μέικ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν με πειράζει που με χαρακτηρίσατε λόμπιστ, αλλά να προσπαθήσω να απαντήσω τώρα στην ουσία της παρεμβάσεώς σας. Εγώ δεν μίλησα για το θέμα της ουδετερότητας του δικτύου, μίλησα όμως για την διακανονιστική αυτή ε, σχέση ανάμεσα στις, στους κατασκευαστές τηλεπικοινωνικών συστημάτων και τους παρόχους και τους υπόλοιπους. Εγώ δεν πρεσβεύω ότι κάθε φορά, αυτός, ε, κάθε φορά θα πρέπει να υπάρξει μια ρύθμιση η οποία να αναγνωρίζει το κεντρικό ρόλο του παρόχου ας πούμε ή κάποιας κυρίαρχης πλευράς αλλά θα πρέπει και σε επίπεδο ευρωπαϊκό, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε επίπεδο εθνικό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η κατάσταση του ανταγωνισμού ανάμεσα στους υπάρχοντες παίκτες, τους λειτουργούντες παίκτες. Και θα πρέπει έτσι να δούμε ποια είναι η επίδοση την οποία έχουν όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό ο τομέας αυτός λειτουργεί στον ανταγωνισμό και σε σωστές ρυθμίσεις και διακανονισμούς. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να απαλλαγούμε από τους διακανονισμούς και τις ρυθμίσεις, αυτό θα ήταν γελίο. Και δεν θα εξυπηρετούσε κανόν, κανένα, θα ήταν παράλογο. Υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα ε, με τα δεδομένα σαν παράδειγμα που αυξάνονται συνεχώς. Πρέπει να επενδύσουμε για να αντιμετωπίσουμε την αύξηση αυτή επενδύουμε. Καλό θα ήταν όμως ε, οι συνθήκες ε, να ήταν ευκολότερες από ό,τι είναι αυτές που παρουσιάζονται σήμερα. Οι ελλείψεις ε, των επενδύσεων, γιατί υπάρχουν τόσες λίγες επενδύσεις, είναι περίπλοκη η απάντηση και δεν μπορεί να δοθεί μια απλή απάντηση όπως η έλλειψη ενιαίας αγοράς. Και αυτό παίζει ρόλο, αλλά είναι ένα τμήμα του προβλήματος μόνο. Και να έρθω στην ερώτηση του Μάλκολμ ε, για τις ε, συμβάσεις και τους όρους των συμβάσεων. Αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα να είχα πει είναι ότι υπάρχουν επιχειρήσεις ε, γύρω από την Ευρώπη και μέσα στην Ευρώπη, μία από αυτές είναι η Deutsche Telekom, που είναι έτοιμες να μεταφέρουν συμβάσεις για μεγαλύτερη διάρκεια από 24 ώρες. θα πρέπει τα ευρωπαϊκά όργανα αν θέλουν να ζητήσουν έτσι ώστε η Deutsche Telekom να επενδύσει περισσότερο χρήμα ε, και να περάσει από τον αριθμό ημερών που είναι σήμερα στη μία ημέρα. Αλλά λαμβάνοντας υπόψη κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες θα βλάψουν τον καταναλωτή Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει γιατί μπορεί να προκαλέσει ακόμα και διακοπές στην παροχή της υπηρεσίας. Η κυρία Μπράνταλ. Να αναφερθώ σε ένα σχόλιο που ακούστηκε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θα έπρεπε να μπορούν να κάνουν καινοτομία στο διαδίκτυο. Σωστό αυτό, αλλά μην ξεχνάμε κάτι. Δεν μπορούμε να θεωρούμε δεδομένο το διαδίκτυο. Υπάρχουν πολλέ εταιρείε που πρέπει να επενδύσουν για να υπάρχει δυνατότητα του διαδικτύου, να υπάρχει κατάλληλη ταχύτητα και κατανάλωση για να καλύπτουν οι ανάγκε μα. Πρέπει αυτέ οι εταιρείε να βλέπουν ότι υπάρχουν κέρδη όσον αφορά που αποκομίζουν τι επενδύσει του. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Συζητήσαμε τους γενικούς κανόνες για την προστασία των καταναλωτών. Και τώρα περνάμε στο δεύτερο πάνελ. Εν τω μεταξύ έφτασε και συνάδελφος Μπάστος, θα της δώσω το λόγο στο τέλος αφού κάνουν τις παρεμβάσεις τους οι φιλοξενούμενοι. Πρέπει να συζητήσουμε τώρα την καινοτομία. Ταυτόχρονα εγγυόμενοι την πρόσβαση στο δίκτυο και προστατεύοντα τα δικαιώματα των καταναλωτών. Μια ουδετερότητα του δικτύου που θα πρέπει να είναι εγγυημένη πρώτος που θα μιλήσει στο δεύτερο τμήμα των εργασιών μας. Eh, Να δώσω το λόγο αμέσως στην κυρία Νάντια Τραϊνάρ της Άρτσεπ που κατέφθασε. Παρακαλώ και εσείς δέκα λεπτά που είχαν όλοι οι υπόλοιποι μετά από σας θα μιλήσει ο κύριος Τσέπερσεν. Λοιπόν, κυρία Τράινερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να εκπροσωπήσω την Μπέρεκ και να σας πω ποια είναι η ανάλυση που έχουμε κάνει και ποια είναι η εμπειρία μας όσον αφορά τη διαμόρφωση πολιτικών και πιο συγκεκριμένα ποια είναι η εμπειρία της Μπέρεκ. Είμαι από τη Γαλλική Ρυθμιστική Αρχή. Εκπροσωπώ την Μπέρεκ σήμερα άρα θα μιλήσω αγγλικά και ζητώ συγγνώμη για, από τους Γάλλους συναδέλφους θα μιλήσω αγγλικά παρότι Γαλλίδα η, η ανάλυση μας όσον αφορά την δετερότητα ε, μας κόστησε με πολλές προσπάθειες το εξετάζουμε το θέμα το 2009 έχω μια σύντομη διαφάνεια που σας δείχνω Ελπίζω να μην είμαι εμπειρογνώμων που θα είναι ενοχλητικός. Έχω μόνο τέσσερις διαφάνειες και προσπαθώ να σεβαστώ το δεκάλεπτο. Η πρώτη πρόκριση για την ΠΕΡΕΚ ήταν να καταλάβουμε καλύτερα τι συμβαίνει στο δίκτυο, να βοηθήσουμε ο κόσμο να καταλάβει τι συμβαίνει στο δίκτυο, σε κάποιο βαθμό να ηρεμήσουμε τι συζητήσει και να υπάρξει καλύτερη επαφή μεταξύ του κόσμου του διαδικτύου και του κόσμου των τηλεπικοινωνιών. Αυτό ήταν ο πρώτο σκοπό. Θέλαμε να καταλάβουμε γιατί είναι σημαντικό για του εμπορευόμενου, για του εμπλεκόμενου, Γιατί έχει σημασία η οδετερότητα του δικτύου Υπάρχει ευρύ φάσμα πρακτικών που ακολουθούνται σήμερα που θα μπορούσαν να υπάρχουν και θα υπάρξουν στο δίκτυο. Κάποιες πρακτικές είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των δικτύων, κάποιες μας έδειξε οικονομική ανάλυση ότι ίσως δημιουργούν προβλήματα στην καινοτομία μακροπρόθεσμα. Η όλη αξιολόγηση της κατάστασης, κυρίως η διαχείριση της κυκλοφορίας ήταν αντικείμενο έρευνας που κάνει το 2012 και έδειξε ότι η κατάσταση δεν ήταν απελπιστική ούτε επιδεινωνόταν. Ο κίνδυνος είναι σημαντικός αν επιδεινωθεί η κατάσταση όσον αφορά την ουδετερότητα. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Δεύτερο στάδιο. Από τις διάφορες πρακτικές που ακολουθούνται Θέλαμε να δούμε ποιες αρχές θα θέλαμε να ακολουθεί η αγορά. Και έτσι προβάλαμε κάποιες αρχές για να αξιολογήσουμε τη διαχείριση της κυκλοφορίας, αν είναι λογική, αν υπάρχουν κριτήρια. Διότι η διαχείριση της κίνησης, της κυκλοφορίας και όλοι οι, συμβα... οι συμβασιακοί μάλλον περιορισμοί, η αντιμετώπιση της κυκλοφορίας ε, αντιμετωπίζονται ποικιλόμορφα. Κάποιε πρακτικέ που ακολουθούνται δεν απαραίτητα επιβλαβεί, χρειαζόμαστε κάποιε έννοιε για να τι αναλύσουμε. Τονίζω και αναφέρω τα κριτήρια, κάποια από τα κριτήρια, διότι πιστεύουμε ότι κάποια από τα κριτήρια ίσω να βοηθήσουν τη βελτίωση, στη βελτίωση των κειμένων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο έλεγχο του τελικού χρήστη, παραδείγματο χάρη, και η προτίμηση ε, για τον αγνωστικισμό όσον αφορά τι εφαρμογέ τι θεωρούμε σαν καλές αρχές που πρέπει να ακολουθηθούν από αγοράς. Θέλαμε να δούμε αυτό και τι μπορούν να κάνουν οι ρυθμιστικές αρχές. Κινηθήκαμε στο διαθέσιμο πλαίσιο, δηλαδή οδηγίες του 2009. Πρώτα απ' όλα, για να προστατεύσουμε την βετερότητα, θεωρήσαμε ότι είναι να λειτουργήσουν οι δυνάμεις της αγοράς, να είναι ανταγωνιστική αγορά να υπάρχει αποτελεσματική διαφάνεια. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και αυτή είναι από τις πρώτε κατευθυντήριες γραμμέ τη Μπέρεκ. Και σωστά λέτε ότι υπήρχαν κάποιες διατάξεις στο πλαίσιο που ίσως δεν εφαρμόστηκαν επιτυχώς και πλήρως. Παραδεχόμαστε ότι ίσως όλα αυτά να μην αρκούν. Ακόμα και μία εύρυθμα λειτουργούσα αγορά, ίσως μακροπρόθεσμα να έχουμε προβλήματα με τη ουδετερότητα. Γι' αυτό είπαμε ότι χρειαζόμαστε ενεργή παρακολούθηση. Να παρακολουθούμε την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται, να βλέπουμε πώς εξελίσσεται η αγορά. Τρίτον, πρέπει να μπορούμε, αν χρειαστεί, να δράσουμε. Αν δεν κάνουμε κάτι τέτοιο, καταστρέφουμε την εμπιστοσύνη των ε, πολιτών. Δηλαδή πρέπει οι πολίτες να πιστεύουν ότι αν υπάρξουν προβλήματα έχουμε εργαλεία παρέμβασης. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αρχές διαλειτουργικότητας, διαδευθετήσεις των διαφορών ή απαιτήσει για ελάχιστη ποιότητα των υπηρεσιών που ήταν ένα από τα νέα εργαλεία που προσέφερε το νομοθετικό πλαίσιο. Αυτά κάναμε λοιπόν με το ισχύον πακέτο. Τώρα με τον νέο κανονισμό τι γίνεται. Έχω αυτή την αστεία διαφάνεια που βλέπετε να σας υπενθυμίσω ότι όλα αυτά εντάσσονται σε ένα πλαίσιο ζωηρής, πολύ ζωηρής συζήτησης τα τελευταία χρόνια. Εδώ παρουσιάζουμε σημαντικά τις προτάσεις για την ουδετερότητα του δικτύου που είναι κάτι επίμαχος διότι δεν υπάρχει επιθυμία δημόσιας παρέμβασης στο διαδίκτυο. Από την άλλη πλευρά όμως ζητείται δημόσια παρέμβαση για την προστασία του διαδικτύου. Κυρίως να προστατευθεί το διαδίκτυο από τους εμπορευόμενους φορείς. Και αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν δικές ιστορίες. Λένε ότι αυξάνεται η κυκλοφορία και δεν έχουν τον άλογο κέρδος και αυτό είναι σημαντικό επιχείρημα που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αυτό είναι το πλαίσιο λοιπόν. Η επιλογή της ρύθμισης του κανονισμού θέτει διαφορετικό πλαίσιο από το παλιό αυτός ο κανονισμός από ό,τι παλιό. Ήταν πιο ήπια η νομοθεσία. Η, πα... Ε, παλιά ίσως σύσταση θα μπορούσε να θεωρηθεί το πλαίσιο του οποίου κινούμαστε. Αν τώρα έχουμε στα χέρια μας κανονισμό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πώς θα συνταχθεί ο κανονισμός διότι το περιβάλλον αλλάζει πολύ γρήγορα. Η Μπέρεκ πιστεύει ότι η πρώτη πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής πετυχαίνει μια αρκετά καλή ισορροπία. Αυτή είναι καλή αρχή. Σχεδόν με ντροπή μου λέω, το λέω αυτό, διότι η Μπέρεκ έχει πολλές επιφυλάξεις για το κείμενο αυτό και ίσως να είναι ίσως εδώ να είναι ο μόνος τομέας ε, που είμαστε ικανοποιημένοι για τον τρόπο προσέγγισης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πώς χρησιμοποιήσετε τα πορίσματα της Μπέρεκ Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια, θα έχω κάποια πράγματα να πω, θα σα απογοητεύσω. Έχω δύο διαφάνειες με βασικά ζητήματα που θα ήθελα να τονίσω. Θα μπω σε τεχνικέ λεπτομέρειε τώρα και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα πρέπει να καθορίσουμε τι υπηρεσίε πρόσβαση στο διαδίκτυο και τι εξειδικευμένε υπηρεσίε. Υπήρχε αυτή η επιλογή στο κείμενο για του ορισμού. Πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμοι ορισμοί. Πολλοί συζητούνται αυτές, αυτοί οι ορισμοί. Θα είναι μάλλον ατέρμονη συζήτηση. Σε κάποια φάση πρέπει να αποφασίσουμε. Πιθανότατα θα ήταν καλό, χρήσιμο. Οι ορισμοί δεν θα πρέπει να είναι πολύ περιορισμένοι για την υπηρεσία πρόσβαση στο διαδίκτυο να ισχύουν οι κανόνες ε, για την αγορά. Ταυτόχρονα οι εξειδικευμένες υπηρεσίες μπορούν να διευκρινιστούν περαιτέρω διότι μάλιστα κάτι τέτοιο θα μας βοηθούσε στην αξιολόγηση της συνύπαρξης εξειδικευμένων υπηρεσιών και υπηρεσίας πρόσβαση στο διαδίκτυο. Εάν εμφανίζεται συγκεκριμένα το πώς εφαρμόζονται αυτές οι αρχές τότε θα μπορούμε να αξιολογήσουμε τη διάδραση μεταξύ των αρχών και να δούμε κατά πόσο στο διαδίκτυο επιδεινώνεται. Πιστεύουμε λοιπόν ότι πρέπει να έχουμε αρχές που θα μας βοηθούν όσον αφορά τα εμπόδια για την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Εμπόδια, αν είναι ακριβή η υπηρεσία που προσφέρεται, η πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά δεν ξέρουμε ποιε θα είναι εξειδικευμένε υπηρεσίε αύριο. Κάποιε από εμά ξέρουμε σήμερα. Παράδειγμα, ε, τηλεόραση μέσω διαδικτύου, μέσω, παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου. Ε, αύριο μπορεί να υπάρχει διαφορετική διάδραση με το διαδίκτυο. Άρα χρειάζεται ευελιξία για να προβλέψουμε μελλοντικέ εξελίξει. Δεύτερο θέμα, οι κανόνες που θα πρέπει να διέπουν την υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο. Σαν Μπέρεκ με χαρά βλέπουμε ότι κάποια σημαντικά για μας κριτήρια συμπεριλαμβάνονται και πάλι. Κάτι σημαντικό που θέλουμε να πούμε. Η αξιολόγηση των πρακτικών. Οι αρχές για προβληματισμό περί πρακτικών που αναφέρονται είναι σωστές. Δεν πρέπει όμως να βλέπουμε μόνο πρακτική εφαρμογή στα δίκτυα αν υπάρχει μπλοκάρισμα ή συμφόρηση της κυκλοφορίας. Δεν λέω ότι είναι χθεσινό πρόβλημα, διότι έχουμε σε κάποιες αγορές αυτό το πρόβλημα ακόμα. Ίσως αύριο να υποβόσκει περισσότερο το πρόβλημα, να μιλάμε για διαφοροποίηση ορίων δεδομένων και καμιά φορά όροι που δεν εφαρμόζονται τεχνικά, αλλά μόνο αναφέρονται στις συμβάσεις. Για τον τελικό χρήστη δεν κάνει διαφορά γιατί δεσμεύεται το περιεχόμενο του συμβολέου. Άρα είναι σημαντικό να έχουμε μια πιο ευρία προσέγγιση στο, στο ζήτημα. Μετά για λογική διαχείριση της κυκλοφορίας των δεδομένων, το δύσκολο ερώτημα είναι ο στόχος. Ποιος είναι? Ο στόχος είναι σχετικός. Υπάρχει ένας κατάλογος στην πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Η προσέγγιση που ακολουθήκε για τον κατάλογο δεν ήταν αυτός της Μπέρεκ, δεν ήταν αυτή της Μπέρεκ. Καλό είναι να υπάρχει κατάλογος, πρέπει να βελτιωθεί όμως ο κατάλογος, διότι υπάρχουν κάποιε κάποιες ασαφείς έννοιες στον κατάλογο και πιθανότατα ο κατάλογος δεν πρέπει να είναι εξαντλητικός. Δεν ξέρουμε ποιε θα είναι οι ανάγκες οι αυριανές για τη λογική διαχείριση κυκλοφορίας. Πρέπει να υπάρχει περιθώριο ελιγμών για τους ρυθμιστικούς φορές, ίσως για την ΠΕΡΕΚ να ξεκαθαρίζουν αυτά τα περίπλοκα ζητήματα που αλλάζουν πολύ γρήγορα. Τελευταία διαφάνεια επιστρέφω στην ελευθερία του ελικού χρήστου σε αυτή την έννοια, διότι συζητήθηκε εκτενώς. Αναφέρεται ότι τώρα όχι μόνο προωθούμε την πρόσβαση του, του χρήστου στο περιεχόμενο, πρέπει να εξασφαλίζεται αυτή η πρόσβαση. Σαν ρυθμιστική αρχή καταλαβαίνουμε ότι οι πολίτες, οι καταναλωτές θέλουν να ωφεληθούν από ισχυρότερη προστασία σχετικά με αυτό το ζήτημα. Θεωρούμε ότι είναι καλό να αναφέρονται οι αρχές Πρέπει να έχουμε ευρύ φάσμα αρχών που αναφέρονται, κάθε είδους κυκλοφορία να καλύπτεται, χρήση τερματικών κλπ. Ταυτόχρονα είναι σημαντικό το κείμενο λαμβάνει υπόψη το ότι αυτή η πρόσβαση στο περιεχόμενο δεν εξαρτάται μόνο από ε, τις εταιρείες, τους παρόχους. Η ιδιαιτερότητα του δικτύου αφορά αυτό που κάνουν οι εταιρείε, ε, οι εμπορευόμενοι στο διαδίκτυο σημαντική πτυχή της χρήσης του διαδικτύου, αλλά η αρμοδιότητα των θυμιστικών αρχών, ο έλεγχος των παρόχων υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, ε, όλα αυτά έχουν κάποια όρια και πρέπει να το έχουμε υπόψη αυτό και να το προσέξουμε. Πιο συγκεκριμένα θέλουμε οι χρήστες να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο και σε εφαρμογές ποιότητας, κάποιες ποιότητας. Πρέπει να έχουμε μια λογική ερμηνεία της έννοιας ποιότητα. Η υπηρεσία πρόσβασης ε, της, ε, στο διαδίκτυο είναι μια υπηρεσία της βέλτιστης προσπαθίας. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να δείξουμε ότι η ερμηνεία του δικαιώματος πρέπει να είναι λογική. Τώρα, για πλευρά του τελικού χρήστη εκεί που έχουμε αρμοδιότητα εμεί αριθμιστικέ αρχές τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να βελτιώσουμε τη διαφάνεια, να σχεδιάσουμε τις μετρήσεις τι ποιοτικέ, να έχουμε συγκρίσιμε μετρήσεις και κάποια ρυθμιστική αρχή στο εθνικό πλαίσιο ίσως να μην έχει όλες τι αρμοδιότητες που απαιτείται και αυτό είναι ένα πρόβλημα προ επίλυση. Υπάρχουν άλλα ζητήματα όμω, όπως η ποικιλομορφία η πολιτιστική, η πολιτισμική ε, και οι περισσότερε μεθυστικέ αρχέ δεν είναι διανοητικά εξοπλισμένε να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα. Λυπούμε που το λέω αυτό. Ε, εγώ είμαι ε, τεχνικό. Και τέλος, η ευρωπαϊκή προσέγγιση είναι πραγματικά σημαντική στο θέμα που συζητούμε. Θα χρειαστούμε η μεν τους δε για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τις περίπλοκες καταστάσεις. Ταυτόχρονα πρέπει να προσέξουμε, δεν θέλουμε αυτό να γίνει εμπόδιο, να μην εμποδίζει μια ρυθμιστική αρχή να κινηθεί και να δράσει γρήγορα με τα διαθέσιμα εργαλεία, τα ενδεδειγμένα εργαλεία, όταν υπάρχει μια προβληματική κατάσταση, διότι το διαδίκτυο κινείται τάχιστα και προσπαθούμε να προσαρμοστούμε δεόντως και να γίνουμε ταχύτεροι ρυθμιστές. Αλλά αυτό είναι ήδη μια πρόκληση. Αυτά εν είδη εισαγωγής. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο κύριο Τζέψεν του Κέντρου για τη Δημοκρατία και Τεχνολογία. Παρακαλώ να σεβαστείτε το χρόνο που έχετε στη διάθεσή μας γιατί έχουμε κάποιους χρονικούς περιορισμούς. Υπάρχει ανάγκη επιτάχυνσης λοιπόν. Ωραία. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για την πρόσκληση να προσέλθουμε εδώ. Η CDT είναι μια ε, εκπρόσωπο τη κοινωνία των πολιτών, μη κυβερνητική οργάνωση. Εργαζόμαστε υπέρ του ανοιχτού και ελεύθερου διαδίκτυου. Ο τίτλος για τη συζήτηση είναι λοιπόν καλά επιλεγμένος, καλά, επελέγει. Και το φόρουμ αυτό, ε, το βήμα αυτό και αυτό σωστά επελέγει, διότι βρίσκεται στην εντολή αυτής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προστασία Συμφερόντων των Καταναλωτών και Προαγωγή της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Εσωτερικής Αγοράς. Δεδομένων αυτών των στόχων, η αμεροληψία και ουδετερότητα στο διαδίκτυο είναι ουσιώδους χαρακτήρα καθορίζοντας τις αρχές ώστε όλες οι νόμιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από το διαδίκτυο δίκτυο πρέπει ίσα και χωρίς διακριτική μεταχείριση να διαβιβάζονται άσχετα από το περιεχόμενο ή τον αποδέκτη. Συνιστούμε λοιπόν σε σχέση με την νομοθεσία για αυτό το επίπεδο ότι είναι ένα καλό επίπεδο, καλό κείμενο, καλή θετική αφετηρία αφήνει όμως και κάποια παράθυρα ανοιχτά που πρέπει να κλείσουν και να ρυθμιστούν. Πρώτα απ' όλα, γιατί η αμεροληψία, η ουδετερότητα στο διαδίκτυο είναι τόσο σημαντική. Και θέλω να το α, τονίσω αυτό. Λένε ότι το διαδίκτυο λέγεται έκανε τεράστια συνεισφορά στην καινοτομία και την ανάπτυξη των οικονομιών μας και έγινε κέριο στοιχείο της καθημερινής ζωής των περισσότερων πολιτών. Πολλά από αυτή την επιτυχία οφείλονται στον ανοιχτό χαρακτήρα του διαδικτύου ως πλατφόρμας, χωρίς περιορισμούς για να υπάρξει ε, ανανέωση της καινοτομίας. Ιδιαίτερα στις εφαρμογές. Το ανοιχτό διαδίκτυο έχει κέρια σημασία και υπό την καινοτομία από πλευρά των επιχειρήσεων και από πλευρά των καταναλωτών. Για τις επιχειρήσεις, τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νεοεισαγόμενες επιχειρήσεις στην αγορά, η ουδετερότητα του διαδικτύου συνολικά σημαίνει ότι εφόσον θα πληρώνει για τη σύνδεσή της μια τέτοια εταιρεία, μια εταιρεία θα μπορεί άμεσα να έχει πρόσβαση στο σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς. Για τις εφαρμογές της υπηρεσίες θα πρέπει να, μπορούν να, να, μπορείτε, να, μπορεί να δημιουργείται ανταγωνισμός έναντι μεγαλύτερων σε μια ανοιχτή οικονομία, σε μια ανοιχτή κοινωνία. Εμείς να ελέγχουμε, εμείς οι πολίτες να αποφασίζουμε ποιες υπηρεσίες, ποιες εφαρμογές θέλουμε να χρησιμοποιούμε, ποιο περιεχόμενο θα διαβιβάζεται, ποιοι θα είναι οι αποδέκτες και με ποιους θα συναλλασσόμαστε διαδικτυακά. Όλα αυτά είναι θεμελιώδη θεμελιώδου σημασία για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε μια δημοκρατική κοινωνία. Η σύνδεση στο διαδίκτυο είναι μια πύλη, η μόνη πύλη σε σχέση με την παγκόσμια διαδικτύωση. Καμιά δημόσια αρχή, η κρατική αρχή δεν πρέπει να είναι σε θέση να περιορίζει ή να ελέγχει και να επιβάλλει επιλογές για λογαριασμό σας. Ε, κάποιοι πάροχοι θα ήθελαν να αλλάξουν αυτά τα πράγματα και να αποκτήσουν διαφορετικό πλαίσιο σύμφωνα με το δικό τους όραμα για το πώς θα πρέπει να λειτουργεί το διαδίκτυο και σίγουρα θα συζητήσουμε περαιτέρω επ' αυτού αργότερα, υστερότερα. Λοιπόν, Όσον αφορά το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες και την προτίμηση αντιμετώπισης ε, ε, στις υπηρεσίες και να πληρώνει κάποιος για προτεραιότητα, αν μετακινηθεί το διαδίκτυο σε μια κατάσταση όπου κάθε ISP θα καθορίζει πώς, υπό ποιου όρους και πόσο γοργά θα μπορούν να έχουν τέτοια συμβόλαια και υπηρεσίες οι καταναλωτές, θα έχουμε ένα πολύ πιο δυσχερές περιβάλλον, πολύ πιο περιεριστικό περιβάλλον. κάθε ε, ε, φορά θα πρέπει να ανησυχεί κανείς τι θα γίνει με τις ISP στις υπόλοιπες χώρες. Και αν σε σχέση με το περιεχόμενο και τις εφαρμογές ε, όλοι εμπλακούν σε αυτό το πλαίσιο, όποιος δεν θα υπογράφει, δεν θα προσυπογράφει μια τέτοια συμφωνία, ένα τέτοιο συμβόλαιο, θα βρίσκεται σε μειονεκτική θέση. Οι γιγαντιές, μεγάλες ε, ε, εταιρείε τηλεπικοινωνιών θα είναι εκείνες οι οποίες θα υποφελούνται και οι μικροί είναι εκείνοι οι οποίοι θα έχουν τις επιζήμες επιπτώσεις. Αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη σε σχέση με τις ρυθμίσεις που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτά τα πλαίσια. Για τα σενάρια, για το ανοιχτό και ελεύθερο διαδίκτυο, με όλα τα ωφέλη για τα οποία ε, έγινε λόγος πιο πριν, να δούμε και το σενάριο όπου οι ISP θα, έχουν, ε, θα επιβάλλουν τέλη και πρόσθετα, ε, πρόσθετες ε, εισφορές σε σχέση με τους χρήστες. Θα πρέπει όμως να δούμε ότι αν πρέπει να διασφαλιστεί το ανοιχτό διαδίκτυο και οι ανοιχτές υπηρεσίες θα πρέπει να συμφωνήσετε ότι είναι δικαιολογημένο να καθοριστεί νομικά η ουδετερότητα και η αμεροληψία στο διαδίκτυο ως αρχή που θα διασφαλίζεται. Έχουν γίνει έρευνες σε αυτό το θέμα σε ευρύ πλαίσιο και βρέθηκε ότι σε σχέση με τους χρήστες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν περιορισμούς ε, ή όρους ε, που δεν δίνουν τη δυνατότητα να προαθούν υπηρεσίες. Επίσης βρέθηκαν τεράστιες διακοιμάνσεις και διαφορές από χώρα σε χώρα και υπό το πρίσμα της ενιαίας εσωτερικής αγοράς και το ρυθμιστικό πλαίσιο οι παρεμβάσεις δικαιολογούνται λοιπόν για να αποκατασταθεί το ορθό πλαίσιο. Λοιπόν, είναι σωστό ότι υποβάλλεται πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διορθωθούν τα πράγματα σε μια σωστή ισορροπία. Σημαντικές βελτιώσεις πρέπει να γίνουν και το πιο σημαντικό είναι το κείμενο θα πρέπει αναμφίσιμα και σαφώς να λέει ότι η μη διακριτική μεταχείριση θα είναι η κύρια προσδοκία και η κύρια αρχή άσχετα από την πηγή, το περιεχόμενο των αποδέκτη ε, ε, διαβιβάσεων ε, μηνυμάτων. Θα πρέπει λοιπόν εδώ το θέμα της αρνητικής διακριτικής μεταχείρισης σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών να ληφθεί υπόψη και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη επίσης αναμφίσιμα το θέμα της θετικής διακριτικής μεταχείρισης. Σενάρια όπου το περιεχόμενο και οι παροχές υπηρεσιών θα πληρώνουν για προτιμητέα αντιμετώπιση όπως να μπορεί να αποφεύγει κανείς το να περιμένει στη σειρά μέχρι ότου να εξυπηρετηθεί μετά από άλλους και να έχει προ, προτιμησιακή μεταχείριση. Και έτσι τα ωφέλη του ανοιχτού δικτύου δεν θα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και θα, ε, θα πρέπει να διασφαλιστεί η δυνατότητα <clears throat> να ε, τα έσοδα να ε, έχουν την πηγή μέσα από ένα διαφοροποιημένο πλαίσιο πακέτων υπηρεσιών στους πελάτες με διαφορετικές επιλογές, διαφορετικές τιμές, διαφορετικές ταχύτητες, διαφορετικό όγκο μεταβίβασης ε, δεδομένων και σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ διαδικτυακών υπηρεσιών και εξειδικευμένων υπηρεσιών. Αυτή θα ήταν η σωστότερη προσέγγιση. Θα πρέπει έτσι να διασφαλιστεί ο ανοιχτός χαρακτήρας στο διαδίκτυο για τις υπηρεσίες που είναι αναγκαίο να γίνει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτές οι υπηρεσίες ε, ε, διαχρονικά και σε σχέση με τον ρόλο που πρέπει να ε, αναλάβουμε επιτηρώντας την κατάσταση των πραγμάτων αυτό έχει κέρια σημασία. Άσχετα πόσο καλά θα μπορέσουμε να καθορίσουμε τη, τους όρους ε, είναι τα πράγματα υποεξέλιξη στις αγορές και θα πρέπει αυτές τις εξελίξεις και τις αγορές να επιτηρούμε. Επαρκούμε σε αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Ανδρέα Ρέντα από το ΤΣΕΠΣ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα σας μεταφέρω τις απόψεις μου για ένα θέμα αρκετά περίπλοκο θα έλεγα. Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι είναι θετικό το ότι συζητάμε αυτή τη στιγμή το θέμα της ουδετερότητας του δικτύου. Πριν 6-7 χρόνια στις Βρυξέλλες αυτό που πίστευαν ότι ούτε η εσωτερική αγορά ούτε το διαδίκτυο θα μπορούσε να είναι πρόβλημα για την Ευρώπη. Όλοι πίστευαν ότι θα υπάρξει μια εσωτερική αγορά για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και δεν είχε δημιουργηθεί πρόβλημα και στις Ηνωμένε Πολιτείε μετά από την απόφαση Madison River. Γιατί στην Ευρώπη εμείς επειδή έχουμε ανταγωνισμό περισσότερο τα λοιπά δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Δεν είναι έτσι πλέον τα πράγματα και συζητάμε τώρα τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της ουδετερότητας του δικτύου. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι μιλάμε για το 2016, 17, 18 Πρέπει να στραφούμε στο μέλλον δηλαδή όταν προετοιμάζουμε τις προτάσεις μας. Και είμαι βέβαιος ότι πολλοί από εμά γνωρίζουν ότι οι τεχνολογίες θα έχουν αλλάξει πάρα πολύ από σήμερα μέχρι το 2017. Σκεφτείτε πριν, πριν πέντε χρόνια ο πιο πολλής κόσμος δεν είχε έξυπνα κινητά τηλέφωνα, smartphones. Ο τρόπος με τον οποίο μπαίνουν οι επιχειρήσεις επίσης και χρησιμοποιούν το διαδίκτυο είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό με αυτό που γινόταν πριν πέντε χρόνια. Τα πρώτα τρία λεπτά της παρουσίασής μου λοιπόν θα δείξουν ακριβώς το τι σημαίνει η ιδέα της ρύθμισης. Το πώς εσείς θα μπορούσατε να τεκμηριώσετε τη διατύπωση ενός κανονισμού στο συγκεκριμένο τομέα. Θα πρέπει να ξεκινήσετε αναγνωρίζοντας ότι μέχρι τώρα έχει υπάρξει μια σχετική αποτυχία των ηγετικών επιχειρήσεων να καθορίσουν τους κανόνες λειτουργίας. Σαν ευρωπαϊκά όργανα και σαν ρυθμιστές θα πρέπει να αναγνωρίσετε ότι η σχεδίαση του αρχικού πακέτου 2002 και 2009 αναθεωρημένο δεν οδήγησε τελικά σε, μια πραγματική εσωτερική αγορά για τις τηλεπικοινωνίες. Εγώ διαφωνώ με αυτούς που πιστεύουν ότι αυτό είναι κάτι το μακροπρόθεσμο, αλλά συμφωνώ με αυτούς που ε, λέγουν ότι η ενιαία αγορά είναι το απτό αποτέλεσμα, το τελικό προϊόν, η είσοδος στις νέες αγορές. Η δυνατότητα συμμετοχής ε, επιχειρήσεων από διάφορες χώρες να φτάνουν στους πολίτες ακόμα και σε επίπεδο ε, λεπτομέρειας. Λοιπόν, δεν μπορούμε εμείς να μιλάμε απλά για μια σύγκληση ε, εποπτικών διαδικασιών. Και γι' αυτό θα περίμενα στις αιτιολογικές σχέσεις του κανονισμού ή στην μελέτη επιπτώσεων να υπάρξει αναγνώριση του ότι οι κανόνες τους οποίους ε, μέχρι τώρα σεβαστήκαμε δεν είχαν σχεδιαστεί για να πετύχουμε την ενιαία αγορά, αλλά για να απελευθερώσουν τις εθνικές αγορές που ήταν περίκλειστες από τα εθνικά του σύνορα. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές ερμηνείες του ότι υπάρχει τεράστια ανάγκη από επενδύσεις δικτύων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ανάγκη ακριβώς επενδύσεις και σε χωρητικότητα δεν είναι μόνο για τη βελτίωση των υποδομών στις τηλεπικοινωνίες, αλλά όλες οι ε, υποδομές που χρησιμοποιούμε σήμερα στον τομέα του ηλεκτρισμού, της ενέργειας κτλ. θα πρέπει να συγκλίνουν στο επίπεδο της ε, τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών τα επόμενα χρόνια. Ε, Εφηή δίκτυα, σαν παράδειγμα, διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και πάρα πολλές άλλες εφαρμογές εισαγωγικά που απαιτούν ε, μια σωστή σύγκληση η οποία να είναι ανθεκτική, συνεχώς λειτουργούσα, υψηλότατα αποδοτική. Αυτός είναι ο στόχος και είναι δύσκολος να τον πετύχουμε. Εδώ ίσως υπάρχει μια κάποια αποτυχία διακανονιστική έχουμε αποτύχει κάτι σε σχέση ε, με το οποίο θα πιστεύαμε ότι ο στόχος μας ήταν ακριβώς μια καθολικά παρεχόμενη υπηρεσία. Οι κανόνες του 09 για τη διαφάνεια βέβαια δεν είναι εύκολο να εφαρμοστούν στην πρακτική. Ο, ο παρακαθήμενος εδώ έδειξε ακριβώς το περίπλοκο χαρακτήρα της δουλειάς των εθνικών εποπτικών αρχών και ακριβώς η ασφάλεια χρήσης του δικτύου είναι κάτι το οποίο σημαίνει διαφορετικά πράγματα για κάθε χρήστη. Θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς απαιτήσει υπάρχουν σε επίπεδο μικροδιαχείρισης της αγοράς και αυτό ε, αποδεικνύει αν θέλετε το ότι βρισκόμαστε σε μια σχετικά δύσκολη κατάσταση σήμερα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε επίσης ότι δεν μπορούμε να πρεσβεύουμε την ουδετερότητα του δικτύου από το 1980 και 90. Ε, πάρα πολύ συχνά ακούγεται ότι ε, έτσι και αλλιώ το διαδίκτυο είναι κάτι το οποίο λειτουργεί με αναρχικό τρόπο. Είναι κάτι στο οποίο ο καθένας τελικά κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να ελέγξει κανείς το ότι κάνει η NSA σαν παράδειγμα και ακόμα και ένας γενικός εισαγγελέας ε, έχει πει στα πλαίσια μιας δικαστικής διαδικασίας ε, ότι ίσως να κληθούν σε κάποια φάση οι πάροχοι να κλείσουν ε, τις ιστοσελίδες οι οποίες διακινούν πειρατικά κλεψίτυπα προϊόντα. Συνεπώς λοιπόν εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι να ζητήσουμε από τις δημόσιες αρχές να ελέγξουν το ίντερνετ. Υπάρχει κάτι το παράδοξο σε αυτή την πρόταση και το οποίο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε. Στο όνομα της ε, ε, ουδετερότητας ε, του διαδικτύου ζητάμε έναν σκληρότατο και αυστηρότατο έλεγχο της λειτουργίας του διαδικτύου. Για να διασφαλίσουμε δηλαδή το επίπεδο της ελευθερίας και της έλλειψης διακρίσεων δημιουργούμε ένα σύστημα παρακολούθησης σε καθημερινή βάση. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε αυτά τα οποία λέω μέχρι τώρα. Πιστεύω όμως ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει κάποια θετικά στοιχεία και ο τρόπος με τον οποίο επεξεργάζεται το θέμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρουσιάζει μια θετική πλευρά και μια αρνητική πλευρά. Η θετική είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαφωνήσει κανείς ότι μπορούμε να έχουμε ένα ανοιχτό ίντερνετ και εξειδικευμένες ε, πάνω από αυτό υπηρεσίες. Από την άλλη όμως εδώ ξεκινάνε τα προβλήματα. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε καταρχάς ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί συγκεκριμένη πρόταση στην πρακτική. Αυτό σημαίνει μία μόνιμη περιπολία σε όλα τα επίπεδα για συγκεκριμένες ε, εφαρμογές και, σας, και για συγκεκριμένους κωδικούς ZIP στο σύνολο του διαδικτύου. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Απ' την άλλη θα αρχίσουμε να συλλέγουμε δεδομένα, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε έναν έλεγχο του διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο. Στα δύο λεπτά τα οποία μου μένουν θα ήθελα να διασφαλίσω ότι τα μέλη του Κοινοβουλίου πρέπει να αποφύγουν τρία διαφορετικά σύνδρομα τα οποία συνδέω με τη συγκεκριμένη πρόταση. Η το πρώτο σύνδρομο είναι το σύνδρομο Γκαλιλαίο. Σε ποιο βαθμό μπορείτε να ε, προτείνετε μια τρομερή υποδομή, μια νέα υποδομή, να ζητήσετε από τον ιδιωτικό τομέα να πάρει μέρο στην υποδομή αυτή, αλλά να του πείτε στον ιδιωτικό τομέα, κοιτάξτε, εμπορική εκμετάλλευση καπούτ. Λοιπόν, ε, στην ουσία θυμάστε τι έγινε, Μάλκομ ξέρεις πολύ καλά με τον Γαλιλαίο, χρειάστηκε να τριπλασιαστεί η δημόσια ευρωπαϊκή επένδυση γιατί δεν υπήρχε ιδιωτική συμμετοχή λόγω της έλλειψης εμπορικών ευκαιριών. Λοιπόν, στις Ηνωμένε Πολιτείε ξέρετε ακριβώς τι γίνεται εκεί με την ουδετερότητα του δικτύου. Άλλο είναι το να είναι κανείς ουδέτερο σε σχέση με τα δεδομένα και άλλο να, να κληθεί να μοιραστεί το δίκτυο με τους ανταγωνιστές του. Ένα άλλο σύνδρομο ε, είναι το να σκεφτούμε ένα δίκτυο ανοιχτό στην πρόσβασή του, ένα άδειο όμως στο εσωτερικό του διαδίκτυο. Το ότι είναι ανοιχτό μπορεί να μειώσει τις δυνατότητες τις οποίες έχει κανείς στο εσωτερικό του διαδικτύου. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ καλό. Σαν να λέμε ότι θέλουμε μια μεγάλη εσωτερική αγορά, ενιαία αγορά, αλλά άδεια στο εσωτερικό της. Όχι. Ε, το θέμα είναι επίσης ένα άλλο σύνδρομο, το σύνδρομο ε, θα έλεγα της υπερβολικής συγκέντρωσης σε ένα συγκεκριμένο χώρο, σε ό,τι φωτίζει η λάμπα της, ε, του δρόμου τη νύχτα. Ε, δεν είναι κάτι τέτοιο πρόθεσή μας. Νομίζω ότι οι τελικοί χρήστες, και αυτά θα τα πει ο Μπελτρά καλύτερα από μένα, έχουν την δυνατότητα μέσω αυτής της αλυσίδας αξιών θα έλεγα, να ζητήσουν την δυνατότητα ελέγχου του διαδικτύου, ε, φιλτραρίσματος του περιεχομένου το οποίο διακινεί ο πάροχος, έτσι ώστε αυτό να βελτιώσει τις εμπειρίες του καταναλωτή πελάτη. Αυτό είναι περισσότερο βέβαια και πρόβλημα εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού και εδώ υπάρχει δυστυχώς πάρα πολύ χώρος για συζήτηση. Ευχαριστώ. Γκουλιέλμου Μπετρά της Μπέου, τελευταίος που θα μιλήσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Χάρμπορ που κάλεσε την Ευρωπαϊκή κατανάλωση, ε, Οργάνωση Καταναλωτών να μιλήσει το σημαντικό θέμα. Για εσά που δεν ξέρετε το BUIC, BOIC, μπορεί να διαλέξετε, προφέρετε την οργάνωσή μα όπω θέλετε. Είμαστε η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών. Εκπροσωπούμε τα συμφέροντα πάνω από 40 εθνικών οργανώσεων ε, καταναλωτών από πάνω 30 χώρε και είναι πρόκληση για μένα να είμαι ο τελευταίο στο πάνελ. Διότι καταρχά, διότι με βάλατε δίπλα μετά με τον κύριο Ράνταλ, που δεν είναι πολύ εύκολο αυτό, σαν ρόλος και επειδή πολλά από τα πράγματα που θα ακούσετε τώρα με κάποιο τρόπο έχουν ήδη αναφερθεί. Σας παρακαλώ να δείξετε υπομονή απέναντί μου. Στην Break Μπέικ λέγαμε ότι το πακέτο 2009 δεν εκάλυπτε παρκώς ε, το ζήτημα, δεν υπήρχαν αρκετά μέτρα διαφύλαξης, ίσως να είμαστε από τους ελάχιστους που λέει ότι ότι από τότε λέγαμε ότι δεν κάναμε αρκετά το 2009 και μας απέδειξε ότι είχαμε δίκιο η ιστορία και χαιρετίζουμε το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας σήκουσε και ανέλαβε σχετική νομοθετική δράση. Η Ρίστον Παρόδο άκουσε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που επανειλημμένως εξέδωσε διάφορα ψηφίσματα και ζητούσε νομοθετική λύση από αυτού όπως και ο κύριος Ράινχαρντ, η κυρία Ράινχαρντ ε, έδειξε διαφάνειες, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Αλλά τάχιστα να διαλύσω κάποιους μύθους ε, που ακούγαμε και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πιστέψουμε στα βασικά στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, επανειλημμένα τέθη το ερώτημα γιατί ζητούμε ρύθμιση του διαδικτύου. Δεν μιλάμε κάτι τέτοιο, δεν μιλάμε κάτι τέτοιο σήμερα. Θέλουμε να ρυθμίσουμε την πρόσβαση στο διαδίκτυο. So, so remain... ώστε διαδίκτυο να παραμείνει ανοιχτό και ουδέτερο. Ο Δεύτερος μύθος ε, που πάντα ακούμε είναι ότι είναι μια λύση που προσπαθεί να βρει πρόβλημα. Ε, δεν είναι αληθεύει, υπάρχει πρόβλημα και πολλοί προλαλήσαντες και μέλη του Κοινοβουλίου συμφωνούν μαζί μας. Τα στοιχεία της Μπέρεκ δείχνουν ότι το 2012 παραδείγματο χάρη ένας από τους τρεις ευρω... κινητής δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει το πρωτόκολλο στα κινητά του VOIP, Voice over Internet και δύο από τους τρεις ε, Ευρωπαίους ήταν αντικείμενο διάκρισης λόγω των παρόχων τηλεπικοινωνιών που εστιαζόταν σε ειδικευμένε υπηρεσίες και αυτό δεν είναι αποδεκτό και νομίζουμε ότι αυτό καθορίζει το πρόβλημα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν στοιχεία, ότι υπάρχει μια τάση τη αγορά για περισσότερες τεχνικές και εμπορικές διακρίσεις. Είτε είναι θετικέ αυτέ είτε αρνητικές. Πιστεύουμε ότι η αγορά δεν θα επιλύσει τα προβλήματα αυτά, αλλά χρειαζόμαστε νέους κανόνε για το παιχνίδι. Οι διακρίσει αυτέ στην πρόσβαση του διαδικτύου, είτε είναι θετικέ αυτέ είτε αρνητικέ τεχνική οικονομική φύσεω, μειώνουν την επιλογή του καταναλωτή και εμποδίζουν την καινοτομία. Ακριβώ επειδή δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η νέα εφαρμογή στο διαδίκτυο, δεν μπορεί στα χέρια τη εταιρεία να αποφασίσει τι επιτυχεί και τι μη επιτυχεί ιδέε. Παράδειγμα τεχνική διακρίση ίσω να είναι ένας, ε, μια εταιρεία που καθιστά σχεδόν ανέφικτη να χρησιμοποιήσει κανεί το WhatsApp ή το Skype. Όλοι συμφωνούμε ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Ε, η οικονομική διάκριση θα ήταν εταιρεία που τιμολογεί διαφορετικά ανάλογα με το περιεχόμενο που αποφασίζω εγώ να χρησιμοποιήσω από τη σύνδεσή μου στο διαδίκτυο. Και όπω ο Γέν ανέφερε προηγουμένω, συμφωνούμε, δεν βλέπουμε πώ η πρόταση αυτή αντιμετωπίζει το θέμα και τα ίδια είδη διακρίσεων είναι, ε, δημιουργούν προβλήματα ή πρέπει να ρυθμιστούν. Εντάχει να αναφερθώ στο τι σημαίνουν αυτά τα δικαιώματα για τον καταναλωτή. Κατά την άποψή μα, να το πούμε απλά, αυτό το δικαίωμα σημαίνει ότι ο καταναλωτής πάντα είναι εκείνο που επιλέγει το περιεχόμενο, υπηρεσίε, εφαρμογέ Μπορεί να χρησιμοποιήσει μέσω του διαδικτύου ε, με ισότιμη αντιμετώπιση. Και αυτό το δικαίωμα πρέπει να προστατευτεί. Για μας αυτό είναι ζήτημα προσδοκιών του καταναλωτού. Το διαδίκτυο από όταν δημιουργήθηκε πάντα ήταν κάτι εύκολο να χρησιμοποιήσει ο πολίτης. Δηλαδή μπορούσε να συνδεθεί και να το χρησιμοποιήσει. Κανείς δεν είχε αμφιβολία πότε ένα νέο πρωτόκολλο ή μια εφαρμογή θα λειτουργούσε στο διαδίκτυο. Πάντα υποτίθεται ότι λειτουργούσε η εφαρμογή στο διαδίκτυο. Τώρα όλο και περισσότερο αυτό εξαρτάται από το, την εταιρεία που σου παρέχει την υπηρεσία του διαδικτύου, την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα τώρα, όσον αφορά την πρόταση που έχουμε μπροστά μα, πιστεύουμε ότι οι καταναλωτέ χρειάζονται αυτό το δικαίωμα, όχι ελευθερία, δικαίωμα. Δηλαδή, όταν έχουν συνάπτων σύμβαση που χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε εξοπλισμό του διαδίκτυο για περιεχόμενο και εφαρμογέ χωρί περιορισμό κανέναν. Εκτό από όρια ταχύτητα και ίσω ε, όρια όγκου. Αν το σκεφτείτε και ένα όριο ταχύτητα ήδη είναι και ένα όριο όγκου. Μετά πρέπει να πείτε στι εταιρείε που πρέπει να σέβονται αυτό το δικαίωμα. Εξαιρέσει από τη γενική απαγόρευση να χρησιμοποιήσουν τη διαχείριση τη κυκλοφορία ίσω θα έπρεπε να προβλέπετε, αλλά πρέπει να αναφέρετε σαφώ στη σύμβαση, μάλλον σε νομοθετικό μέτρο. Η συμμόρφωση με τι εντολέ του Δικαστηρίου για την ασφάλεια του διαδικτύου κατά επιθέσεων, η μείωση των αποτελεσμάτων προσωρινών και εξαιρετικών περιπτώσεων συμφόρηση είναι λόγοι για τη διαχείριση των δικτύων, νόμιμοι, αλλά πρέπει να αναφέρονται ε, σαφώ και να προβλέπονται. Συμφωνούμε με την προσέγγιση τη Μπέρεκ, δηλαδή προσέγγιση με βάση τον κατάλογο. Νομίζω ότι είναι σωστή. Επίση, να μην λησμονούμε ότι οι κατανοτέ στην Ολλανδία και τη Σλοβενία έχουν αυτά τα δικαιώματα προστατευμένα ισχυρά. Εφόσον είναι ένα κανονισμό αυτό που θα οδηγήσει σε μέγιστη εναρμόνιση, θα ήταν απαράδεκτο αν αυτοί οι καταναλωτέ χάσουν ε, κάποιο δικαίωμα. Για εξειδικευμένε υπηρεσίε, αν νομιμοποιηθούν και αριθμιστούν όπω αυτή είναι η πρόθεση, τότε χρειάζονται μέτρα διαφύλαξη ισχυρή για να προφυλάξουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τι σχετικέ υπηρεσίε. Δυστυχώ, οι προτάσει που έχουμε δει σχετικά με αυτό είναι αόριστες και μπορεί να οδηγήσουν σε κενά. Θα πρέπει να ενισχυθούν. Θέλω επίσης να θέσω δύο ερωτήματα για τις ειδικευμένε υπηρεσίες. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα για υψηλής ποιότητας συνδετησιμότητας δεν εμποδίζουν την ποιότητα της πρόσβασης στο διαδίκτυο στους καταναλωτές. Μέχρι στο αναλυθεί όλο αυτό, το άρθρο 19 της πρότασης θα πρέπει να διαγραφεί. Δεύτερον, για τις εξειδικευμένες υπηρεσίες. Στο βαθμό που εξειδικευμένες υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται πάντα, θα πρέπει οι εταιρείε να έχουν κίνητρα για να, έχουν, να περιορίζουν το εύρος που διαθέτουν. Πώ θέλουμε να σίγουρα ότι οι εταιρείε θα επενδύουν για να δημιουργούνται υποδομέ που είναι υπέρ των προϊόντων γενικά του διαδικτύου και όχι για τι εξειδικευμένε υπηρεσίε. Τέλο, να το πω ειλικρινά, παρόλο που τα μηνύματα δεν είναι πάντα σαφή, ο τομέα των επικοινωνιών, τουλάχιστον ένα τμήμα αυτού του τμήματο, δεν θέλει να αφήσει του καταναλωτέ να διαλέγουν τι υπηρεσίε και το περιεχόμενο ισότιμα. Ε, ισότιμα, το τονίζω. Όπω είπε και ο Γιέν, στην πράξη κάποιε εταιρείε θέλουν όλο το διαδίκτυο να λειτουργεί διαφορετικά και να υπάρχουν οι πάροχοι περιεχομένου που θα πληρώνουν αυτού για την παροχή ε, του περιεχομένου, σαν είναι ταχυδρομείο. Δεν είναι 19ο αιώνας, δημιούργησε προσθέμενη αξία το διαδίκτυο, όντα ανοιχτό και φιλικό προς την καινοτομία. Αυτή η νομοθετική μεταρρύθμιση δίνει όλο την ιστορική δυνατότητα να ενισχύσουν και να προστατέσουν το διαδίκτυο για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσουμε το θέμα των ερωτήσεων και απαντήσεων δίνοντας το λόγο αμέσως στην κυρία Μπαστός, η οποία είναι σκιώδης εισηγήτρια για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Έχετε το λόγο κύριε Μπαστός. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ξεκινώ ζητώντας συγγνώμη για την απουσία μου κατά το πρώτο πάνελ. Δεν ήταν δυνατό να είμαι παρούσα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων και έτσι δεν μπόρεσα να παραστώ κατά την έναρξη αυτής της ενδιαφέρουσας συζήτησης στο πρώτο πάνελ. Και συγχαίρω σε αυτό, το δεύτερο πάνελ για τον τρόπο με τον οποίο διαμόρφωσαν τις παρεμβάσεις τους σε ένα τέτοιο ευαίσθητο θέμα όπως την ουδετερότητα στο διαδίκτυο και όσον αφορά τα προϊόντα και τις επιχει... τις... Ε, την παροχή υπηρεσιών την ισορροπία που πρέπει να διασφαλιστεί μεταξύ υπηρεσιών ε, που θα παρέχονται επιχειρήσεων και καταναλωτών και όσον αφορά το πακέτο Telecom αυτό το θέμα της ουδετερότητας του δικτύου διαδικτύου ήταν εκείνο που Σα απασχόλησε περισσότερο. Φυσικά από τότε μέχρι σήμερα υπήρχε μια δυναμική ανάπτυξη, μια εξέλιξη πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι παρόλες τις προσπάθειες των νομοθετών να παρακολουθήσουν τα πράγματα στις τηλεπικοινωνίες ε, έχουμε μπροστά μας ε, ορόσημα και προκλήσεις και συμφωνούμε ότι οι αρχές που πρέπει να διέπουν αυτό το θέμα της ουδετερότητας στο δίκτυο είναι αρχές που πρέπει να είναι υγιείς και στερεές και πρέπει να συμφωνήσουμε ότι θα είναι αρχές που πρέπει να προσαρμόζονται σε αυτό το δυναμισμό, δυναμική εξέλιξη του τομέα και δεν πρέπει να παρακολύουν νέες υπηρεσίες και νέα προϊόντα που θέλουν να εισέρχονται στην αγορά Υπό αυτό το πρίσμα θα πρέπει οι υπηρεσίες να μπορούν να, να η παροχή υπηρεσιών να προβλέπουν δυνατότητες εξυπηρέτησης των καταναλωτών, των χρηστών. Ένας τρόπος να εξευρεθεί αυτή η ισορροπία θα ήταν να καθορίσουμε με σαφήνεια μια διαχωριστική γραμμή, τη διαχείριση τεχνική της, δια, της των μηνυμάτων σύμφωνα με σαφείς όρους ε, που θα διέπουν αυτό τον τομέα αφενός και αφετέρου την διαχείριση του εμπορικού, των εμπορικών, εμπορικών συναλλαγών <clears throat> που αν δεν γίνει αυτό μπορεί να υπάρχουν καταχρήσεις. Γι' αυτό το θέμα μου, η ερώτησή μου προς τους ε, πραγματογνώμονες που παρενέβησαν σε αυτό το δεύτερο πάνελ. Η ερώτησή μου, τι θεωρείτε, πώς θεωρείτε αυτή τη διαφοροποίηση μεταξύ τεχνικής διαχείρισης ε, των κανονικών συναλλαγών και των εμπορικών συναλλαγών. Με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να καθορίσουμε σαφώς και την μεν και την δε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι θέλουν να μιλήσουν. Κυρία Βερχόιεν. Και εγώ από πλευράς μου θέλω να ζητήσω συγγνώμη που ήρθα με κάποια καθυστέρηση σχεδόν στο δεύτερο πάνελ. Ταυτόχρονα είχαμε μια σε βάθος έντονη συζήτηση στην Επιτροπή Πολιτισμού που αφορούσε και γνωμοδότηση για την ε, ενιαία εσωτερική αγορά ε, τηλεπικοινωνιών και το περιεχόμενο αυτό και έπρεπε να, ήμουν, να είμαι παρούσα εκεί γιατί είμαι σκιώδη εισηγήτρια γι' αυτό. Καταρχήν θέλω να πω την προσέγγιση που εδώ εν μέρη παρουσιάστηκε από πλευρά των εισηγητών σε σχέση με την ακρόαση την υποστηρίζουμε και πάλι την ε, προσέγγιση του εισηγητή σε πολλούς τομείς δηλαδή σε σχέση με την οδηγία να μπορέσουν κάποια πράγματα να διαγραφούν επειδή υπάρχουν πρωτοβουλίες ε, ήδη νομοθετικά πλαίσια έχουμε το πακέτο 2009 για τις τηλεπικοινωνίες που εγκρίθηκε που το 2011 εν μέρη υλοποιήθηκε σε κάποια κράτη-μέλη αν κιόλα υλοποιήθηκε και σε όλα και πολλά σημεία αναφέρονται εδώ και πιστεύω ότι ε, μέσω Μπάρακ έχουμε ένα θεσμικό όργανο, ένα θεσμό που ας το πω έτσι τον έλεγχο συγκεκριμένων τομέων ή την παρατήρηση, την εποπτεία συγκεκριμένων τομέων σε, με καλό θετικό αναλυτικό τρόπο έχει παρουσιάσει και πολλές προτάσεις μπορούν να είναι εφικτές. Για το θέμα της ουδετερότητας του δικτύου φυσικά δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο τους ίδιους τους καταναλωτές. Το θέμα της ουδετερότητας του δικτύου είναι αφορά και το περιεχόμενο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη δημιουργική, δημιουργική ευφυή παραγωγική οικονομία. Πολύ σημαντική αυτή η προσέγγιση. Θα με ενδιαφέρε συγκεκριμένα εδώ και πάλι πώς η εισαγωγή νέων υπηρεσιών νέων υπηρεσιών υπό το πρίσμα της διαχείρισής τους, διασφάλιση ποιότητας, εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπως και να τις αποκαλέσουμε, ποιες επιπτώσεις θα έχουν όλα αυτά στις μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, που σε μια πολύ ανταγωνιστική πλευρά των τηλεπικοινωνιών, ως επιχειρήσεις ε, εξαρτώνται από την υψηλή ποιότητα της διαβίβασης και χρειάζονται ένα ανοιχτό διαδίκτυο και εξαρτώνται ενδεχόμενα και από εξειδικευμένες ε, υπηρεσίες. Όταν έχουμε εκατοντάδες ε, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών που αγωνίζονται για να κλείσουν συμβάσεις και συμβόλαια με χρήστες και όταν έχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες αν ξεχωριστά αντιμετωπιστούν σε μια δομή στο δίκτυο δεν κάνω λόγο για την υποδομή των δικτύων γιατί τα ίδια τι τις ίδιες υποδομές χρησιμοποιούν τα δίκτυα, αλλά πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε νέες υπηρεσίες να μπορούν να εισαχθούν, που ταυτόχρονα με την εκμετάλλευση των υποδομών και την διεύρυνση των υποδομών δεν θα αποβαίνουν εις βάρος ενός ανοιχτού δικτύου ή εις βάρος της ποιότητας. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Βερνιού. Πολύ γρήγορα θέλω να συγχαρώ το δεύτερο πάνελ. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για μένα τουλάχιστον. Αντιστοιχούσαν αυτά που είπαν στις ερωτήσεις που έθετα. Πιο συγκεκριμένα βεβαίως το θέμα της ουδετερότητας του δικτύου. Πράγματι κάποιος αναφέρθηκε στα προηγούμενα χρόνια και στο πακέτο τηλεπικοινωνιών του 2009. Νομίζω ότι οι χρήσεις ήταν διαφορετικές και εξελίχθηκαν ταχύστα και θα εξελιχθούν πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε στεναροί όσον αφορά το μπλοκάρισμα των υπηρεσιών καθώς και τις υποχρεώσεις περί διαφανείας. Και πραγματικά σχεδόν σε όλα, και αυτό δεν με εκπλήσει, σχεδόν σε όλα συμφωνώ με την παρέμβαση ε, της Μπέρκ που θέτει το θέμα, το πρόβλημα. Πώς θα εγγυηθούμε το δικαίωμα του καταναλωτού να επιλέγει ανεφορείων χωρίς διακρίσεις. Αυτό μπορεί να θέσει κανείς σαν θέμα περισσότερων δικαιωμάτων και σε ποιο επίπεδο θα γίνει εναρμόνιση για να μην χαθούν δικαιώματα. Αυτό εννοούσα και στην αρχή. Βέβαια, θα χρειαστεί να επαγρυπνούμε τα μάλλα όσον αφορά τη διαχείριση της ε, κίνησης, της και την διακριτική πρόσβαση. Ε, θα πρέπει να προχωρήσουμε στο μέτρο του δυνατού με τη βοήθεια ειδικών σίγουρα των παρόντων όσον αφορά τον ορισμό των εξειδικευμένων υπηρεσιών ή των κλειστών δικτύων λαμβάνοντας ε, υπόψη όλες τις διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των διαφόρων ειδών υπηρεσιών και των διαφόρων ειδών δικτύων. Σε αυτό ε, μας διαφωτίσατε και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τη συνέχεια του προβληματισμού και σας ευχαριστώ για αυτό. Ευχαριστώ. Άγκστρομ. Κύριος Άγκστρομ. Ευχαριστώ. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπα για το προηγούμενο πάνελ. Ευχαριστώ τους συμμετέχοντες σε αυτό το πάνελ. Κυρίως τον εκπρόσωπο της οργάνωσης ε, των καταναλωτών. Συμφωνώ, είναι ένα πρόβλημα του πραγματικού κόσμου. Πράγματι επηρεάζει άμεσα τους καταναλωτές και συμφωνώ με κύριο Βερχόιεν, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η δυνατότητα νέων προσφορών, όπως είπε η κυρία Βερχόγεν, όχι μόνο από μια χούφτα εταιριών τηλεπικοινωνιών σε κάθε εταιρεία, αλλά εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που πράγματι είναι η ρεχοκοκαλιά της ευρωπαϊκή οικονομίας. Και πρέπει αυτές να έχουν ασφαλές περιβάλλον για να μπορούν να έχουν πρόσβαση ε, στο διαδίκτυο με τους ίδιους όρους που έχουν και όλοι οι άλλοι. Ευχαριστώ. Ο εισηγητής πρόεδρος έχει το λόγο, κ. Χάρμπορ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλη την ομάδα. Νομίζω ήταν πολύτιμη η παρέμβασή τους. αφαιθώ σε κάποια θέματα που αντιμετωπίζουμε. Δεν θα σας εκπλήσει δεδομένου του περιεχομένου της πρότασης που σας δόθηκε ότι βασιστήκαμε κατά πολύ στην πολύ καλή δουλειά της Μπέρεκ. Αναφέρθηκε αυτό. Είχαμε συμπεριλάβει ιδιαίτερα όρους. Θέλαμε να δούμε τι τι σημαίνει εμπόδιο και επιδείνωση της πρόσβασης ε, στο διαδίκτυο και μιλώ ποιότητα, ε, τιμή ε, και άλλους παραγόντες που βάζουν την πρόσβαση. Δηλαδή, πώς μπορούν και οι ρυθμιστικές αρχές να κινηθούν βάσει αυτών. Ο Άντριου Ρέντερ ή κάποιος άλλος μίλησε για την διάκριση με, λόγω τιμών. Σωστά αναφέρθηκε αυτό. Υπάρχουν διάφοροι τομείς διάκρισης. Δεύτερον, με ενδιαφέρουν οι εξειδικευμένε υπηρεσίε. Είναι νέο ορισμό. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο Κρίστιαν Έγκστρομ νωρίτερα. Οι υπηρεσίε βίντεο δεν είναι ιδιαίτερα καλό παράδειγμα εξειδικευμένων υπηρεσιών, διότι δεν χρειάζονται τόσο μεγάλη ε, ποιότητα. Είναι αρκετά καλή η ταχύτητα τώρα με τα νέα πρωτόκολλα του διαδικτύου. Τα ακούσαμε και το πρωί μα, το είπε ειδικό. Το ερώτημα είναι τι είναι εξειδικευμένε υπηρεσίε. Τι θα είναι. Στην αρχή δεν ήμουν σίγουρος ότι έπρεπε να εφεύρουμε νέες υπηρεσίε. Παρόλο που κάποιοι αυτό υποστηρίζουν. Αυτό πίστευα αρχικά αλλά μου είπε η Μπέρεκ ότι δύο στους τρεις Ευρωπαίους ε, υποφέρουν διότι ε, γίνονται κείμενο διάκρισης λέω ότι εστιάζονται οι εταιρείε στις εξειδικευμένες υπηρεσίες. Θέλω να ξέρω ακριβώς τι είναι αυτές οι εξειδικευμένες υπηρεσίες και τα στοιχεία που προέρχονται. Αυτό θέλω να μου πει η Μπέρεκ. Δεν είδα εγώ τέτοια στοιχεία πουθενά ούτε κι άλλοι συνάδελφοι εδώ δεν ξέρω πως συνάδελφοι θεωρούν ότι αντικείμενο διάκρισης λόγω εστίασης στις εξειδικευμένες υπηρεσίε. ούτε δύο στους τρεις από το ακροατήριο θέλω να ξέρω περισσότερα και ίσως από αυτό θα συναγάγουμε ε, συμπεράσματα τι πρέπει να κάνουμε και κάτι άλλο που δεν εφήγει αλλά ίσως θα θέλαμε το σχολείο συμπέρι θα το πω τώρα Πρέπει να δράσουμε τώρα. Είμαι αγνωστικιστή στην προσέγγιση μου. Η Μπέρεκε έχει ασχοληθεί με το θέμα, έχει εξουσίες για την ποιότητα και τη διαφάνεια. Αλλά βλέπω ότι οι κυβερνήσεις σε διάφορες χώρες της Ευρώπης με αυθαίρετο τρόπο θεσπίζουν δικές τους ρυθμίσεις για την ουδετερότητα του διαδικτύου αυτό θα οδηγήσει σε κατακαιρματισμό της αγοράς. Πρέπει να διατηρήσουμε ένα κοινό πλαίσιο για να παίρνουν αποφάσεις επενδυτές. Γι' αυτό είμαι υπέρ του κανονισμού για ανοιχτή πρόσβαση στο διαδίκτυο, για να έχουμε ένα συνεπές πλαίσιο. Τα απόγευμα άκουσα με ενδιαφέρον ότι η Ολλανδική κυβέρνηση μάλλον θα εγκρίνει κάποια νομοθεσία σχετική είδαν τι πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είπαν δεν είναι αρκετά τολμηρό, αρκετά καλό και θα θεσπίσουν νέα νομοθεσία στην Ολλανδία. Αν κανεί ξέρει κάτι παραπάνω, α το αναφέρει. Πριν ολοκληρώσουμε το νομοθέτημα, α δούμε τι κείμενα έχουν περάσει σε άλλε χώρε. Η ομάδα μου των ειδικών το εξετάζει αυτό και το εξέτασε και γι' αυτό καταλήξαμε σε σχετικέ τροπολογίε. Θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. και προσπαθήσαμε από την υπάρχουσα τεχνογνωσία να αντλήσουμε γνώσεις και να προτείνουμε κάποια πράγματα. Αυτά ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ζητώ από τους φιλοξενούμενους μας στην ίδια σειρά που ακολούθησαν για να μιλήσουν να απαντήσουν στις τεθήσεις ερωτήσεις για ένα δίλεπτο ο καθής. Η κυρία Τράινερ ξεκινήσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Απλά ίσως σύντομα για να επανέλθω στο θέμα, στις παρατηρήσεις της κυρίας Βερνιό, σε ερωτήσεις της. Πώς να συνδέσουμε το θέμα των τεχνικών. Η κυρία Μπάστος το ρώτησε. Τεχνικές πτυχές και εμπορικές πτυχές, εμπορικούς όρους. Το 2009 είπαμε, εκθέσαμε ότι οι ίδιες αρχές μπορούν για τις σταθερές και τις κινητές επικοινωνίες να εφαρμόζονται. Αυτή η αρχή για την οποία κάνουμε λόγο τώρα εφαρμόζεται και στις τεχνικές και στις εμπορικές ε, χρήσεις. Ε, ε, δεν χρειάζεται να έχουμε διαφορετικές αρχές να χρησιμοποιήσουμε. Μια από τις αρχές είναι ο έλεγχος ε, τελικών χρηστών. Ακούμε για διάφορα επίπεδα όπου ο προβληματισμός λέει μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε το κείμενο για την επιλογή χρηστών. Κάτι άλλο που αισθάνομαι υποχρεωμένη να αναφέρω, γιατί δεν υπάρχουν άλλοι εκπρόσωποι από το πάνελ, <clears throat> για το θέμα της, ε, συμβατότη, ε, ε, συμβατότητας και ουδετερότητας όσον αφορά τις χρήσεις και εφαρμογές μεταξύ χρηστών, παρόχων υπηρεσιών και ITTs το να έχουμε συγκεκριμένες τέτοιες αρχές σημαίνει ότι θα πρέπει συγκεκριμένες εφαρμογές να προσφέρονται. Δεν είναι μόνο η προσφορά του διαδικτύου με, ε, διάφορες, ε, με διάφορα πριμ. Πρέπει να δούμε την εξειδικευμένη μορφή των ε, χρήσεων. Πρέπει να υπάρξει μια ευκαιρία να λειτουργήσει αυτό. Αυτό υπονοεί βέβαια ότι θα έχουμε επίσης καθήκον να επιτηρούμε τα όσα θα συμβαίνουν στο διαδίκτυο σε σχέση με αυτά Κατανοώ την ε, ανησυχία προλαλήσαντος ότι η εποπτεία από πλευράς ε, ε, των εποπτικών αρχών δεν είναι ακριβώς εκείνο το οποίο είχαμε εμεί υπόψη. Αλλά η επιτήρηση για να δράσει κανείς είναι καλύτερη επιλογή από το να έχουμε αντιμετώπιση κάποιων περιορισμών μετά από πλευράς προσφορών. Αυτή η, αυτή η προσέγγιση που επελέγει νομίζω είναι η ορθή. Ευχαριστώ. Uh, I Μπορώ uh, να υποστηρίξω σχεδόν όλα όσα η συνάδελφος προανέφερε. Θα έλεγα για τις εξειδικευμένες υπηρεσίες για την, το ερώτημα τι ακριβώς ε, είναι αυτές οι υπηρεσίες που θα απαιτήσουν αυτόν τον ειδικό, ας το πω έτσι, την ειδική αντιμετώπιση, ειδικά επίπεδα παροχής υπηρεσιών ε, που δεν μπορούν να παρασχεθούν ε, μέσω του κανονικού διαδικτύου ως υπηρεσίες. Από πλευράς παρόχων αναφέρθηκε ότι είναι αναγκαίο να μπορούν να παρέχονται αυτές οι υπηρεσίες και να χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να παρισφρέουν στην αγορά και για την εποπτεία δεν είναι απόλυτα σαφές πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και τι θα γίνεται σε σχέση με την δυνατότητα επόπτευσης της κατάστασης. Αυτό θα είναι ένα κέριο θέμα στη συνέχεια. Άσχετα ποιοι ορισμοί θα υιοθετηθούν, πόσο καλά θα διατυπώσουμε τους ορισμούς στον κανονισμό και τα συναφή. Ένα άλλο θέμα το οποίο αναφύεται είναι γιατί γιατί εξετάζουμε το θέμα των διατάξεων για την μη διακριτική μεταχείριση και την ουδετερότητα του δικτύου στη συνολική συζήτηση. Πρέπει να επανέλθω σε αυτό το οποίο αναφέρθηκε. Κάνουμε λόγο για την ανοιχτή πρόσβαση στο δίκτυο. Δεν κάνουμε λόγο για οποιοδήποτε και παντός είδους υπηρεσιών στο διαδίκτυο. Αυτό είναι προσχηματικό και δεν πρέπει να γίνεται. Και τέλος θα ισχυριζόμουν ότι υπό τους όρους ε, της ε, αναλογία ISP ε, και των κυριότερων εμπλεκόμενων πιστεύω ότι αν η δική σας επιχείρηση παρέχει στους πελάτες ανοιχτή πρόσβαση στο διαδίκτυο θα είναι προς το δικό σας συμφέρον να υπάρχει ένα οικοσύστημα εντός εισαγωγικών που θα βοηθά την ανάπτυξη και τις εφαρμογές που θα επιθυμούν οι χρήστες να χρησιμοποιούν. Διότι αυτό είναι που θα δίνει το κίνητρο να, αναβαθμίζουν, ε, να αναβαθμίζονται οι συνδέσεις ε, και να καλύπτονται και τα έξοδα. Ευχαριστώ. Okay, thank you very much. Remarks... Σας ευχαριστώ πολύ κάποιες παρατηρήσεις για τα θέματα που προαναφέρθηκαν, ιδιαίτερα το θέμα της ε, εισόδου και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην πρόσβαση αυτή. Ένα που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι πρέπει να διατηρήσουμε υπόψη ότι όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, φαίνονται σαν να έχουν ένα πολύ μεγάλο εύρος στην μέση και όχι στο, στην κορυφή και στην βάση σε σχέση με τους παρόχους ε, περιεχομένου υπηρεσιών. Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι μια κατάσταση όπου μεγάλο μέρος του δυναμικού ε, ε, παρέχεται από τα, τις διαστρωματώσεις εφαρμογών με πολλά σημαντικά προτερήματα και πλεονεκτήματα. Όμως υπάρχουν πολύ λίγα κίνητρα και προτερήματα για όσους βρίσκονται πάνω-πάνω και κάτω-κάτω σε αυτή την ε, κατακόρυφο, σε αυτόν τον άξονα. Και πρέπει να δούμε τι γίνεται σε σχέση με τις ε, επιχειρήσεις των ΗΠΑ και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Προτού πούμε ότι είναι τεράστιο το επίτευγμα αυτό το οποίο επετεύχθη από εμάς για την πρόσβαση και τις νεοσερχόμενες εταιρείες, ας ξαναπροβληματιστούμε γι' αυτό. Όχι επειδή πιστεύουμε ότι δεν ήταν ε, θετικό επίτευγμα, αλλά επειδή συνολικά η ICT, οι πληροφορίες, η πληροφόρηση και οι τεχνολογίες ε, πληροφορίας ε, δημιουργούν ένα κενό εδώ μεταξύ ΙΠΑ και Ευρώπης. Και για την, τις νέους ερχόμενες θέλω να καταγγείλω τον μύθο για το πώς μπορούν να εισέρχονται οι νέες εταιρείε σήμερα στην αγορά. Υπάρχει διαχείριση των πραγμάτων και ε, σε σχέση με εταιρείε, ε, για παράδειγμα, που έχουν εφαρμογέ ε, για το iPhone, δεν είναι αυτό ένα ανοιχτό δίκτυο. Υπάρχει μια εταιρεία που εκμεταλλεύεται ένα συγκεκριμένο φάσμα με την εκμετάλλευση ιδεών και εφαρμογών. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί τι κάνουμε ο ανοιχτός χαρακτήρας είναι εκείνος που δίνει κίνητρα για να, νέο, να υπάρχει η δυνατότητα νέου εισερχόμενος σε αυτόν τον τομέα. Μία τελική παρατήρηση πιστεύω, αλλά αυτό θα πρέπει σίγουρα να ξανασυζητηθεί γιατί θα υπάρχουν παρεκκλείσμουσες απόψεις. Δεν είναι μόνο προς το συμφέρον των τελικών χρηστών να υπάρχει μη διακριτική μεταχείριση και ανοιχτό χαρακτήρας. Πρέπει να υπάρχει και σωστό μείγμα ε, υπηρεσιών και επιλογών. Επιλογές που είναι σημαντικές βασικό θέμα να μην επιδοτούνται ή ενισχύ, ε, υποστηρίζονται οικονομικά κάποιες υπηρεσίες και απαιτείται μετά η υποστηριζονται οικονομικα καποιες ψηλότερου τέλους για να παρέχονται. Γιατί διαφορετικά αντί για ανοιχτό χαρακτήρα θα οδηγηθούμε σε ομαδοποίηση καταναλωτών σε μία κατηγορία ισοπεδωτικά ενώ θα έχουν τελείως διαφορετικές ανάγκες ημένα από τους δε. Um, Uh, λοιπόν, πάρα πολύ σύντομα θα ήθελα να επανέλθω στην ερώτηση της κυρίας Μπάστος. Αν κατάλαβα καλά, ζήτησε να μάθει τη διάκριση ανάμεσα στη διαχείριση ε, της κυκλοφορίας στο διαδίκτυο για τεχνικούς λόγους ή για εμπορικούς λόγους. Ε, αυτό το οποίο προσπάθησα να εξηγήσω ότι όταν μιλάμε για εμπορικούς λόγους κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να συμβαίνει γιατί αυτό δημιουργεί μια διάκριση. Εάν πράγματι εγώ έχω ε, μια υπηρεσία παροχή στο διαδίκτυο και θέλω να κατεβάσω ε, κάποιο βίντεο ή να επισκεφτώ μια ιστοσελίδα, μια Παρασκευή απόγευμα, ώρα υψηλής χρήσης, θα συμφωνούσαμε ότι θα είναι απαράδεκτο ο παροχέας να περιορίσει ε, πρόσβασή μου ή να διαχειριστεί την ταχύτητα της σύνδεσής μου μόνο και μόνο γιατί έχει υπερβολική ζήτηση στην πλατφόρμα της ψηφιακής τηλεόρασης. Εδώ είναι ένα παράδειγμα στο οποίο η διαχείριση του εμπορικού κομματιού με τη διαχείριση της κυκλοφορίας του δικτύου έρχεται σε σύγκρουση. Φυσικά και απαιτείται μια τεχνική διαχείριση και γι' αυτό όμως ζητάμε μια διευκρίνηση γύρω από το πώς και πότε θα πρέπει να γίνονται όλα αυτά. Οι αριθμοί τους οποίους δίδουμε ε, δίδονται στον έλεγχο των στοιχείων του 2012 για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στο διαδίκτυο. Μπορούμε να σας δώσουμε την ανάλυση της έρευνας αυτής εφόσον το επιθυμείτε. Σας ευχαριστώ. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Βιόλα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά στον εισηγητή για να κλείσει. Ζητώ συγγνώμη εγώ θα πάρω τη θέση του κυρίου Βιόλα, αλλά θα μιλήσω εγώ γιατί δεν ήταν μαζί μας από την αρχή της συζήτησης. Λέγομαι Βίλαν, Γενική Διεύθυνση Connect. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε συγχαίροντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σας και τον εισηγητή σας για την ευκρίνεια με την οποία ολοκληρώνετε τις εργασίες σας Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε μαζί σας και προσβλέπουμε στη στιγμή που το Συμβούλιο θα είναι έτοιμο να κάνει το ίδιο. Γιατί νομίζω ότι αξίζει ε, ε, να γίνει αυτό μετά από την προσπάθεια την οποία έχετε κάνει και το χρόνο που αφιερώσατε σε αυτό το γενικά κατεπήγον θα έλεγα πακέτο. κάτι το οποίο είναι κατεπήγον και για το καλό των εισηγητών ε, και για όλους. Αναφέρθηκα στα δύο αυτά θέματα. Αν δει κανείς καταρχάς ε, το γενικό θέμα της προστασίας του τελικού χρήστη, θα πρέπει να μην αγνοήσουμε όχι μόνο τον στόχο που έχουμε για ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή σε μια, φάση, σε μια αγορά αυστηρά ανταγωνιστική και αποδοτική. Αλλά θέλουμε επίσης να υπάρχει ένα επαρκές πακέτο κοινών κανόνων που θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε σε επιχειρησιακές συναλλαγές μέσω του διαδικτύου ανάμεσα σε όλα τα κράτη. Ε, είναι μια προϋπόθεση αν θέλετε για το τι θα ακολουθήσει. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ακούσαμε τις τρεις διαστάσεις που υπάρχουν, το μέσο, την εναρμόνιση και υπάρχει επίσης και το θέμα της ουσίας του περιεχομένου. Συνδέονται μεταξύ τους αυτά τα τρία επίπεδα. Να αναφερθώ στο περιεχόμενο πρώτα. Να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι αν πράγματι θέλουμε να έχουμε κοινού κανόνες θα πρέπει να βάλουμε το επίπεδο υψηλά, θα πρέπει να υιοθετήσουμε τις πλέον καλές πρακτικές στα διάφορα κράτη-μέλη έτσι ώστε κανένας καταναλωτής να μην είναι σε θέση αδυναμίας. Άκουσα επίσης με προσοχή και τον εκπρόσωπο του Ρίτς, τον κύριο Χούτον, ο οποίος είπε ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία στα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως και εγώ αναγνωρίζω ότι υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία και σε σχέση με την έκθεση την οποία προτείνει ο εισηγητής σας σε πολλούς τομείς. Σύντομα τώρα να έρθω στα άλλα δύο θέματα, στο μέσο και στο επίπεδο εναρμόνισης. Αυτό είναι κάτι το διαφορετικό. Μπορούμε να στοχεύουμε για, σε ένα υψηλό επίπεδο εναρμόνισης μέσω της οδηγίας. Από την άλλη είναι σαφές ότι ένας κανονισμός απαιτεί κοινού κανόνες άμεσα εφαρμόσιμους και άμεσα ε, διαθέσιμους ή τουλάχιστον διαθέσιμους σε μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό είναι κάτι πάνω στα οποία επιμένουμε και σέβομαι εδώ σε σχέση με τις ε, διαφορετικές ίσως ελαφρώς απόψεις της, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του εισηγητή. Θα αναφερθώ στην Πράκνελ σε σχέση με τα μέσα και το υψηλό επίπεδο εναρμόνισης. Νομίζω ότι αν δεν διασφαλίσουμε τις προτεραιότητες αυτές, φοβάμαι ότι ανοίγουμε τους ασκούς του αιώλου για το τι θα ακολουθήσει. Να στραφώ τώρα πάρα πολύ σύντομα στο θέμα της ουδετερότητας του διαδικτύου. Ακολουθώντας τη λογική την οποία μόλις προανέφερα και την ανάγκη ύπαρξης κοινών κανόνων στην εσωτερική αγορά και από, τις δύο, και από τους δύο εισηγητές των αρμόδιων επιτροπών ε, ζητείτε να υπάρξει περισσότερη ε, ρύθμιση. Βέβαια στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα ε, σε κάποιες διαρκείς θα έλεγα χρονικά νομικές ρυθμίσεις και την ανάγκη διαφάνειας και ενιαίου τρόπου εφαρμογής τους στα διάφορα κράτη-μέλη. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύουμε ότι έχουμε επιλέξει τις σωστές αρχές και μπορούμε να προχωρήσουμε στον τομέα της ουδετερότητας. Επί τη βάση της αρχής της μη επιβλαβούς συμπεριφοράς στον τομέα της κυκλοφορίας των δεδομένων κτλ. και της διαφάνειας. Απαιτείται να υπάρξει ένας συγκεκριμένος κατάλογος εγκεκριμένων αποκλήσεων σε αυτές τις βασικές αρχές τις τόσο σημαντικές. Φυσικά και πρέπει να διαφορμόσουμε την δράση μας με συγκεκριμένες αναφορές ε, στους λόγους ύπαρξης, αν θέλετε, της διαχείρισης της κυκλοφορίας των δεδομένων. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι μια υπερβολικά θεωρητική παρουσίαση των α, επιτρεπόμενων αποκλήσεων θα δημιουργήσει προβλήματα και προβληματική γενικά εφαρμογή των γενικών αυτών αρχών. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να σταθώ είναι οι εξειδικευμένες υπηρεσίες. Θα πρέπει να κάνουμε τη διάκριση στο τι είναι και τι δεν είναι, αλλά να αποφύγουμε μια εκ των προτέρων υπερβολική, αν θέλετε, ε, ρύθμιση στον συγκεκριμένο τομέα. το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι και θέμα ας πούμε στον τομέα του ανταγωνισμού. Το δεύτερο θέμα είναι ότι το βασικό τηλεπικοινωνιακό ε, προϊόν είναι η πρόσβαση στο διαδίκτυο. Απαιτούνται συγκεκριμένες αποδείξεις για την ε, απομείωση της σημασίας αν θέλετε ε, της συγκεκριμένης διαδικασίας. Η προτινόμενη νομοθετική ρύθμιση ε, αφορά ε, την κυριαρχία του ανοιχτού ίντερνετ. Ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στις εξειδικευμένες υπηρεσίες, το ίντερνετ πρέπει να μείνει παρα, ε, ανοιχτό και δυναμικό. Υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου των διαδικασιών αυτών για τις τοπικές εποπτικές αρχές οι αρχές αυτές θα είναι σε θέση να δημιουργούν τα ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια έτσι ώστε να διασφαλίζονται ε, τα συμφέροντα των καταναλωτών. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι οι εξειδικευμένες υπηρεσίες θα θα γίνονται αντικείμενο συμβάσεων αν θέλετε μόνο από αυτούς οι οποίοι ειδικά τις χρειάζονται. Εμείς σαν νομοθέτες δεν θα πρέπει να αποφασίσουμε ε, το τι χρειάζεται κανείς για να κατεβάσει ένα βίντεο ή όχι. Αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται εσωτερικά. Εμείς θέλουμε όμως να έχουμε ένα δίκτυο ε, υψηλού επίπεδου χωρητικότητας και ταχύτητας και κανένας χρήστης δεν θέλει να πληρώνει τέλη και προμήθειες για ε, υπηρεσίες τις οποίες δεν χρειάζεται. Και εδώ ο ρόλος των εποπτικών αρχών είναι καθοριστικός. Αυτοί καθορίζουν τους κανόνες. Ε, πιστεύουμε λοιπόν ότι έχουμε την απαιτούμενη βάση για να βελτιώσουμε το κείμενο ακόμα περισσότερο και πάρα πολύ σύντομα να υπάρξει απαιτούμενη σύγκληση σε αυτό το τόσο σημαντικό κοινωνικό αλλά και οικονομικό θέμα. Ευχαριστώ. Ο συγγητής έχει το λόγο για τα τελικά του σχόλια. Ο κύριος Μάκομ Χάρμπορ, το συμπέρασμά μου είναι να ευχαριστήσω πραγματικά όλους τους φιλοξενούμενους επαΐοντες ε, για το ότι αλληλοσυμπληρώθηκαν στα όσα μας είπαν και προσθέθεσαν πολύ χρήσιμες πληροφορίες ε, στα όσα είχαμε. Αυτό δεν διευκολύνει υποχρεωτικά τα πράγματα, αλλά θέλω ιδιαίτερα να πω ότι χαιρόμαστε και οι σκιώδεις εισηγητές ε, και εγώ για το δυνατότητα να προβληματιστούμε επί των σημείων που μας προαναφέρατε. Πέρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα αναφερθώ σε αυτήν σε μια στιγμή, έχουμε εδώ βασικές δομές στη διάθεσή μας. Η βασική δομή που δημιουργείται και τα κυριότερα στοιχεία για το περιεχόμενο αυτών των δομών νομίζω την χάνουν ευρύτερη υποστήριξη. Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες και όπως και η κυρία Τράινερ ανέφερε ε, ο διάβολος πάντα κρύβεται στις λεπτομέρειες σε αυτούς τους τομείς. Θα έλεγα, δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά τα θέματα. Και απαντώντας στην παρέμβαση του κυρίου Βουίλαν, δεν βλέπω κανένα λόγο να υφίσταται. Γιατί οι διατάξεις της οδηγίας που ουσιαστικά στοχεύουν σε ένα στοχευμένο εναρμονισμό όπου τα κράτη-μέλη θα απαιτείται να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν αυτές τις διατάξεις και για τη διάθεση στοιχείων και πληροφοριών. Γιατί θα είναι διαφορετικές από τις διατάξεις που ισχύουν και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Πρώτα, να κατανοηθούν οι υφιστάμενες ε, διατάξεις της υφιστάμενης οδηγίας, υφιστάμενης οδηγίας χωρίς να υπάρχει σύγχυση σε σχέση με μια κεντρική διαχείριση και να λάβουμε υπόψη τις παρεμβάσεις και προτάσεις από πλευρά πλευρά Ευρωκοινοβουλίου και να επιτρέψουμε δεύτερον να προσαρμοστούν και να μετεξελιχθούν και να προχωρήσουν αν χρειάζεται σε σχέση με τις δυνατότητες που θα τους παρασχεθούν στην εφαρμογή όρων και διατάξεων που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν. Ο Άντωνη και εγώ είχαμε ανταλλάξει πολλά επιχειρήματα για όλα αυτά. Αλλά οι συνάδελφοι υποστηρίζουν νομίζω αυτή την προσέγγιση και αυτή είναι η προσέγγιση που θα υιοθετήσουμε. Οι διατάξεις από πλευρά των ρυθμίσεων, η κυρία Τράινερ ήταν ήταν πολύ διπλωματική και δεν το κατονόμασε. Νομίζω και από πλευράς ρυθμιστών ε, υπάρχει ευθυγράμμιση με αυτή την προσέγγιση. Αυτά προτείνουμε εδώ και με την πείρα που υπάρχει σε σχέση με θέματα προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών από πλευράς μας θέλω να υπενθυμίσω ότι εμείς είμαστε εκείνοι που προσθέσαμε συγκεκριμένες αναφορές ε, για να βελτιωθούν τα πράγματα σε σχέση με τις ανάγκες που υπάρχουν σε σχέση με αυτή την οδηγία. Θα λέγα ότι κάναμε πολύ καλή δουλειά για τους καταναλωτές ε, καλύτερη δουλειά από ό,τι έγινε από πλευρά τη αρχική πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμένω και επιμένω σε αυτό. Ελπίζω ότι οι συνάδελφοί μου θα συμφωνήσουν μαζί μου. Θα υπάρξουν φυσικά πρόσθετε διατάξει και ρυθμίσει που θα πρέπει να ακολουθήσουν. Ολοκληρώνω εν τέλει λέγοντα γιατί τέθηκε και το θέμα άλλων πτυχών του συνολικού πακέτου στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις παρατηρήσεις της ε, για την, ε, τις προσπάθειες που έγιναν μέχρι σήμερα και για το τι επετεύχθη. Πρόσθετη αξία πρέπει να δοθεί όσον αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών. Και σε σχέση με το πώς έχουν τα πράγματα, άλλες πτυχές ίσως πρέπει να εξεταστούν από πλευρά των Αν αμένουμε σε σχέση με το τι θα συμβεί με συγκεκριμένες ε, πτυχές και τη μεταξέλιξή τους. Ίσως ε, θα πρέπει λοιπόν να αποφασίσουν οι συνάδελφοι το τι θα πρέπει να γίνει σε σχέση με αυτό. Για την περιαγωγή και άλλες πτυχές όπου έχουμε απόψεις <clears throat> θεώρησα ότι από πλευρά μα δεν θα έπρεπε να υποβληθούν περαιτέρω ε, συστάσει πέρα από αυτέ που, ε, που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή Βιομηχανία. Αν οι συνάδελφοί μου όμω ε, θεωρούν πρέπει να γίνει αυτό είναι ελεύθεροι να το πράξουν. Σα ευχαριστώ όλου λοιπόν για όλα αυτά. Απλά και μόνο να επιβεβαιώσω το χρονοδιάγραμμα επαληθεύοντας κάποια πράγματα. Πρέπει να κινηθούμε ταχύτατα για τι τροπολογίε λόγω του χρονοδιαγράμματο που θεσπίστηκε. Μέχρι τι 3 Δεκεμβρίου πρέπει να έχουν κατατεθεί οι τροπολογίες σα. Θα εξεταστούν προ ψήφιση και έγκριση στι 9 Ιανουαρίου και συμβιβαστικές τροπολογίες στις 22 Ιανουαρίου. Νωρίς το Φεβρουάριο θα ψηφίσουμε. Στις 23 Ιανουαρίου θα συναντηθούμε για να ψηφίσουμε, για να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής ε, Βιομηχανίας. Συμμερίζομαι την άποψη του συναδέλφου Γουίλαν ότι καλό θα ήταν να ξεκινήσουν συζητήσεις με τα κράτη-μέλη αν είναι δυνατόν θα ήθελα να λάβουμε υπόψη σε σχέση με τις συζητήσεις αυτές τις πτυχές για τους καταναλωτές. Δεν θα έπρεπε να ε, υπάρξει κάποια καθυστέρηση ή εμπόδια. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμά μας. Θα δούμε αν θα μπορέσουμε λοιπόν σε σχέση με και τη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών να δώσουμε συνέχεια σε κάποια θέματα με τροπολογίες. Είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε όλες αυτές τις πτυχές. Σας ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον Αντιπρόεδρο, Αντιπρόεδρο και ο Κοφεράτη που προείδρευσε σε αυτή την κοινοβουλευτική επιτροπή μας τώρα, ώστε να μπορέσω εγώ εισηγητής να παρουσιάσω το έργο μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λοιπόν και εγώ και δίνω ξανά την Προεδρία στον uh, κύριο Χάρμπουρ. Αφού ευχαριστήσω και τους φιλοξενούμενους μας.